Um, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me say. Uh, Καλησπέρα. Έχουμε πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα. Επιτάπητος. Το 11 της ημερήσιας διάταξης. Ετικετοθεσία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Επισήμανση τα μέλη έχουν υποβάλει πάνω 500 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Ο Νταρίο Ταμπουράνο είναι εισηγητής. Και είναι η πιο σημαντική έκθεση αυτής της θητείας, η έκθεση του Ντάριο. Λαμβάνει υπόψη την ενεργική απόδοση πολύ σοβαρά και την επισήμανση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη προσέγγιση, ομοιογενής, με σαφείς κανόνες. Για τους πολίτες μας αυτό είναι σημαντικότατο. Λοιπόν, συνάδελφε, Ντάριο Ταμπουράνο, θα μπορούσατε να δώσετε το εναρκτήριο λάκτισμα στη σημαντικότητα αυτή συζήτησή μα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Καλημέρα Μάλλον καλό απόγευμα σε όλους τους παρόντες και σε εκείνους που μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Επιτέλους είμαστε στην πλήρη διαδικασία διαπραγματεύσεων της προτάσεως του κανονισμού όσον αφορά την ετικετασία αυτή την ενεργειακή. δράτα μας ευκαιρίας να ευχαριστώ τους 63 συναδέλφους που υπέβαλαν ή συνυπέγραψαν τις σχεδόν 700 τροπολογίες. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια σημαντική επιβεβαίωση τη βούληση όλων των συναδέλφων να ξεπεράσουν την νομοθετική πρόταση στην αρχική, ενισχύοντά την και εμπλουτίζοντά σε πολλά σημεία. Έναντι μια τέτοια πρώτη ε, εκθέσεω με πολλά σημεία, λάβαμε διάφορε πολλέ ε, αιτήσει για εμβάθυνση. Πάνω από το 1 τέταρτο από τι τροπολογίε Συγγνώμη, είχαμε κάποιο πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρο, ε, όσον αφορά τη διαρμηνία σε κάποιες γλώσσες, όχι σε όλε τις γλώσσες, σε κάποιες γλώσσε, υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Και οι διερμηνείς σας παρακαλούν αν έχετε την καλοσύνη να μιλάτε λίγο πιο αργά. Λίγο πιο αργά, σας παρακαλούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ίσως από την αρχή, λέει ο πρόεδρο. αν, είσαστε, αν έχει την καλοσύνη. Ξεκίναμε και το χρονόμετρο από εκεί. Ορίστε. Καλησπέρα σε όλους τους παρόντες και σε εκείνους που μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Επιτέλους είμαστε στην πλήρη διαδικασία διαπραγματεύσεων της προτάσεως κανονισμού όσον αφορά την ενεργειακή τικητοθεσία και ευχαριστώ τους 63 συναδέλφου που υπέβαλαν ή συνυπέγραψαν σχεδόν 700 τροπολογίες. Πιστεύω αυτό επιβεβαιώνει και με σημαντικό τρόπο τη βούληση όλων των συναδέλφων να ξεπεράσουν τα όρια τη αθλητική νομοθετική προτάσεω, ενισχύοντά την και εμπλουτίζοντά σε πολλά σημεία. Έναντι τη πρώτη εκθέσεώ μα, λάβαμε αιτήσει τροποποίησεω πολύ ενδελεχή και πάνω από τον τέταρτο των υποβληθισών τροπολογιών προσέστησαν ένα κείμενο και δημιούργησε κείμενο εντελώ καινούριο. Το σύνολο των συνεισφορών και πολλέ από αυτέ που επέκριναν μα επέτρεψαν να βελτιώσουμε σημαντικά το κείμενο. Στόχο μα να καταφέρω να συντονίσω τονίσω τι συνεισφορέ σα προ την επεξεργασία μια θέση που αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ε, πλειοψηφία τη Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται από μια σαφή φιλοδοξία που θα είναι απαραίτητη όταν σαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα ξεκινήσουμε τι επαφέ με το Συμβούλιο. Πολλά τμήματα τη προτάσεω ε, είναι αλληλένδετα και θέλουμε να έχουμε μια θέση η οποία να είναι οργανική και να υποστηρίζεται από όλου. Θα ήθελα πολύ η προστασία των πολιτών, η βολή προς το μέλλον και η μείωση των, του άχτους όσον αφορά τις επιχειρήσεις με τη μείωση της χαρτογραφίας, ε, συγγνώμη, της γραφειοκρατίας να βρεθούν τελικά στην τελική λύση. Σας επισημαίνω σε αυτά τα λεπτά που έχω στη διαθεσή μου κάποιες πτυχές σημαντικές. Το μεγαλύτερο ποσό των τροπολογιών βασίζονται στις νευραλγικές πτυχές ε, όσον αφορά το άρθρο 7, τις ετικέθες και την αλλαγή του μεγέθους, κατεξοδότηση πράξης άρθρο 12 και του ορισμούς του άρθρου 2. Οι τροπολογίες όσον αφορά τα 4 άρθρα αντιπροσωπεύουν το 50% εκείνων που έχουν υποβληθεί. Ε, πολλές προτάσεις ευτυχώς είναι δημιουργικές και ακολούθησαν την κατεύθυνση ενίσχυσης τη εποπτείας της αγοράς προς σκοπό να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πετύχουμε την πραγματική εφαρμογή του κανονισμού, άρθρα 5 και 6. Στην ουσία του, το 7 βλέπουμε ότι θα είναι ο συμβιβασμό που είναι αποτέλεσμα συνομιλιών με του συναδέλφου. Δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία, αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δύο προτεραιότητε που πρέπει να εξετάσουμε. Πώ θα συνδέσουμε την διαδικασία του rescaling στην, ε, στις ανάγκες αγοράς και πώς θα τα πετύχουμε αυτά χωρί να αρχίσουμε από την αρχή, να κάνουμε reset την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πραγματιστέ και πραγματικοί χωρί να χάσουμε την, ε, τον όραμά μα. Θέλουμε πολίτε και καταναλωτέ, στου οποίου θέλουμε να δώσουμε εύληπτα σήματα και πλήρη, ούτω ώστε να δώσουμε στο σύστημα τη ετικετοθεσία πλήρη σαφήνεια και αποδοτικότητα. Η ύπαρξη παρα, του κάτι παραπάνω θα καλύψει τα κενά και την, ε, το να μην είναι κατανοητέ οι πληροφορίε. Ε, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τι θα φαίνεται στο σήμα. Λοιπόν, πολλέ ανθρωπολογίε που ζητάνε να υπάρχει βάση δεδομένων. Θα ήθελα να πω ότι αντιθέτω θέλουν να περιοριστούν κάποιε στο πεδίο εφαρμογή ή δεν θεωρούν ότι έχει προτεραιότητα αυτή η εφαρμογή. Όπω ήδη ανέφερα σε άλλε περιπτώσει, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχει πλήρω ο κανονισμό να δημιουργηθεί ένα σύστημα ψηφιακό που θα δώσει πραγματική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι εποπτικέ αρχέ και ταυτόχρονα θα εμπλουτίζει τι πληροφορίε που θα έχει ο πολίτη, ούτω ώστε να μπορεί να ε, εκμεταλλευτεί πλήρω τη δυνατότητα που του δίνει η οικονομία ενέργεια που αναφέρεται στην ετικέτα. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν προσοχή στο κατά πόσο έχουν, ε, πρέπει να προστατεύσουν πληροφορίε βιομηχανικέ που είναι κάπω απόρριτε και ευαίσθητε. Θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα για τη διαφάνεια όπου θα πρέπει να σειραίουν και να είναι προσβάσιμες σε πληροφορίες και έγγραφα που ήδη ε, είναι δημοσίας φύσεως, αλλά είναι δύσκολο να τις βρει κανείς. Είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη βούληση για βελτίωση τη εποπτεία τη αγορά και η διαδικασία τη προστασία για προϊόντα που δεν συμμορφώνονται, έναντι προϊόντων που δεν συμμορφώνονται. Πολλοί συνάδελφοι και σχεδόν όλοι ε, οι ενδιαφερόμενοι συμμερίζονται πολλέ ανησυχίε όσον αφορά την αποδοτικότητα του παρόντο συστήματο εποπτεία. Μια τέτοια πολιτική προσοχή με κάνει να βλέπω με αισιοδοξία τη δυνατότητα να βρούμε μια συμφωνία που θα ε, λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση τη κυκλοφορία των πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών, την βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών, το μεγαλύτερο ρόλο που θα πρέπει να παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συντονισμό αυτών των διαδικασιών στην αγορά τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ήθελα να προσθέσω κάποια άλλα στοιχεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω σήμερα και που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για τη συζήτηση. Θα υπάρχει μεγάλη συνένεση όσον αφορά την ανάγκη αυτό, αυτή η ετικέτα να είναι πολύ ορατή ε, για όποιον πάει στο κατάστημα και σαφώς να βλέπετε η, η ενεργειακή κατανάλωση κάθε προϊόντος. Υπογραμμίζω ότι ο πραγματικός στόχος ε, του κανονισμού ε, λαμβάνοντα υπόψη και τι αποφάσει πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, η μείωση τη ενεργειακή κατανάλωση στο σύνολό τη. Με αυτή την οπτική γωνία, θα πρέπει να επενθυμίσω και να υπογραμμίσω ότι η ενεργειακή απόδοση είναι μόνο το μέσο ούτω ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι μα. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονό ότι υπάρχει αρκετά κοινή προσέγγιση και απέτηση για ενίσχυση των μηχανισμών συμμετοχής και διαβούλευσης και μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εποπτεία της εφαρμογής του κανονισμού. Κλείνω υπογραμμίζοντας την άποψή, που έχει, την άποψή μου για τη σημασία που έχει ε, ε, ε η ψηφιακή, η ψηφιοποίηση των πληροφοριών είναι δυνατότητα να κάνουμε μεγάλο βήμα πρόοδου για την πληροφορία που θα έχει ο πολίτης. Να μειώσουμε το κόστος και το άχθος, ε, που, ε, κάτι που δεν είναι, να είναι καλύτερη και η συσκευασία και να μειώσουμε και την κατανάλωση των φυσικών πόρων, να είναι πιο ελαφριά η συσκευασία. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε ανα οποιαδήποτε στιγμή τις ερωτήσεις που θα αναδειχθούν σε επόμενες μέρες τόσο ώστε η τελική μας θέση να είναι ισορροπημένη και φιλόδοξη, ούτω ώστε να προστατεύσουμε τον καλύτερο τρόπο τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλης της Ένωσης όσον αφορά τα βασικά θέματα της ενεργειακής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο συνάδελφος Ρόιλ έχει το λόγο. Shadow Rapporteur. Ja, thanks. Also, äh, erstens bedanke Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την συνεργασία. Ελπίζω να την ολοκληρώσουμε γέρος. Ε, για μένα το σημαντικό είναι να κάνουμε μια απλή ρύθμιση, να μην έχουμε τίποτα το πολύπλοκο. Λιγότερα πράγματα, αλλά ουσιαστικά. Ουσιαστικά σημαίνει να δημιουργήσουμε ένα μέσο για τον καταναλωτή που θα πετύχει αυτό το οποίο θέμε. Δηλαδή αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. Σημαίνει όμως ότι και yeah. τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους θα πρέπει να είναι το σύστημα λογικό. Και εδώ πέρα υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι η ανακατάταξη. Να προσέξουμε δηλαδή να μην κάνουμε ένα τόσο λεπτομερή κανονισμό που να μην ε, λειτουργεί. Δεν γίνεται να αλλάξουν όλες οι ετικέτες αμέσως. Π.χ. υπάρχουν προϊόντα που άλλαξαν ετικέτες ε, μόλις πέρσι. Δεν γίνεται ε, συνέχεια αυτή η δουλειά. Πρέπει να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε πρέπει να ξανακινηθούμε, να κινείται η Κομισιόν συνεχώς ή όταν ξαναγεμίσουν θα έλεγα, όταν όλες οι συσκευές είναι κατηγορίας Α και Β να συνοηθούμε σε μια προθεσμία η οποία δεν θα είναι μεθαύριο, αλλά να αφήσουμε λίγο χρόνο στους ανθρώπους. Πέντε χρόνια π.χ. Αλλά σημαντικό είναι και το θέμα της τράπεζας δεδομένων. Κάποιοι το βρίσκουν θαυμάσιο, μπορεί, αλλά κοστίζει λεφτά, κόπο και για την Κομισιόν. Αρχαίμε λοιπόν τι νόημα έχει. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Η έκθεση τεστ ενός ε, προϊόντος είναι ολόκληρος χαρτοφύλακας και υπάρχουν ε, εταιρείες που έχουν 10.000 προϊόντα που θα πρέπει να καταγράψουν. Αυτό τι να σου πω, δηλαδή 25.000 προϊόντα, φανταστείτε να το περάσει κανείς σε μια βάση δεδομένων online. Και δεν έχει αποδειχτεί και η αναγκαιότητα. Λέτε τι υπάρχει σε άλλες χώρες, Αυστραλία, ΗΠΑ, Κίνα. Δεν ξέρω, ίσως να έχουν πιο ευέλικτο σύστημα αυτοί από ότι εμάς. Αν δείτε ειδικά ότι εμείς η διαφορά είναι ότι στις χώρες αυτές υπάρχει μία αρχή που ελέγχει μόνο και μία επίσημη γλώσσα. Σε εμάς θα είναι πολλές οι αρχές και οι γλώσσες. Οπότε παρακαλώ να το σκεφτείτε. Η αποτελεσματικότητα της σημερινή ε, κλίμακας είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Ήταν καλή, ας ε, αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες Α, μην τα κάνουμε ακόμη πιο γραφειοκρατικά και δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Για τους σοσιαλδημοκράτες, κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ, η οποία αντικαθιστά την σκιώδη συγγετρία την κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ματίνα δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να είναι εδώ ζητά συγγνώμη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό για τη δουλειά που κάνει. Είναι πολύπλοκος ο κανονισμός, καλύπτει 15 ομάδες προϊόντων, οπότε δυσκολία να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της γενικής και της ειδικής προσέγγισης. Για τις ε, συγκεκριμένες ε, τροπολογίες, το άρθρο 7 είναι η βάση της ε, πρότασης για εμάς είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της αρχικής ανακατάταξης και το να δούμε από ποιο σημείο και μετά θα γίνονται οι μελλοντικές ανακατάταξεις. Εμείς προτείνουμε η αρχική ανακατάταξη να φορά όλα τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εξάλλου ο βασικός στόχος είναι να ξεφύγουμε από την κλάση α3 συν. Εμείς και κάποιες ομάδες έχουμε πει κάποια ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αν δεν ορίσουμε μια σαφή προθεσμία για την αρχική επανακατάταξη, κάποια προϊόντα θα κρατήσουν το α συν συν για 10 χρόνια. Μόλις γίνει αυτό το αρχικό, οποιαδήποτε μεταγενέστερη ανακατάταξη θα πρέπει να γίνει μόνο όταν έχει προχωρήσει επαρκώς η τεχνολογία και οι ανώτερες κατηγορίες έχουν μετά αποκτήσει υπερπληθυσμό. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ένα ποσοστό των προϊόντων που ανήκουν στις δύο κορυφαίες κατηγορίες. Εμείς είμαστε ελεύθεροι, ανοιχτοί να συζητήσουμε ποιο θα πρέπει να είναι αυτό το όριο, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει σταθερότητα και μόλις γίνει η ανακατάταξη να παραμείνουν οι ετικέτες αναλύωτες για 10 χρόνια. Όσον αφορά τις άδειες κατηγορίες όλες οι ομάδες είναι υπέρ ε, είτε της μία είτε και των δύο κορυφαίων ε, κατηγοριών ε, να είναι άδειες. Για εμάς μία ή δύο άδειες για να, μείνουν, για να μην υπάρχει σύγχυση των καταναλωτών, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο καλό συμβασμό με τον εισηγητή και τους κοιόδους. Το ίδιο ισχύει και στο χρόνο που θα δώσουμε για, στους εμπόρους για να αλλάξουν τις ετικέτες. Σχεδόν όλοι έχουν καταθέσει ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα από μια εβδομάδα μέχρι ένα μήνα. Νομίζω μπορούμε χωρίς προβλήματα να συμφωνήσουμε. Για τις πράξεις κατά εφαρμογή και κατά εξοδότηση νομίζω πως η πλειοψηφία είναι υπέρ. Και βεβαίως υπάρχει και η βάση δεδομένων. Γενικά η πλειοψηφία των ομάδων υποστηρίζει την πρόταση της ε, Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το περιεχόμενο και την ε, ουσία και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τώρα λοιπόν περιμένουμε οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές να βρουν ένα καλό συμβασμό που θα στηρίζει η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Γιατί βεβαίως έχουμε και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να έχουμε έναν καλό συμβασμό. Και πάλι ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος της Ματίνας που προψιάζει. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Από το, από το Άλντε, ο Φιλίπ Ντεμπάκ. Εγώ είχα άλλες πληροφορίες ε, ότι θα μιλούσε ο Φρεντερίκ. Όχι, όχι, αλλάζουμε. Ένα παίρνει θέση του άλλου. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Οι συζητήσεις που έχουμε κινούνται με επικοδομητικό τρόπο. Καλό πάντα είναι αυτό. Χθες είδαμε, όταν συζητήσαμε τα άρθρα, ότι μπορέσαμε να βρούμε συμβιβασμού. Αυτό που έχει σημασία για εμάς τους φιλελεύθερους, το έχω αναφέρει και στις παλιές μου παρεμβάσεις, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ετικέτα που ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να μπορούν να, καθα... να καταλαβαίνουν, να είναι πιο ενημερωμένοι και να, κάνουν, ε, να παίρνουν αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως. Επομένως, ακριβώς αυτό θα πρέπει να αντακτοπρίζεται. Το πόσο ε, ενεργειακά αποδοτικό είναι ένα προϊόν. Εδώ μπαίνουν και επισέρχονται πολλά πράγματα και αυτά θα πρέπει να αναφέρει η ετικέτα και αυτά θα πρέπει να δίνει ως πληροφορίες. Δεύτερον, Νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουμε από το παλιό στο καινούριο, όσο πιο ομαλά γίνεται και για τους προμηθευτές και τους παραγωγούς, αλλά και τους εμπόρους. Και, και για μένα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε την αλλαγή στις κλίμακες όπου χρειάζεται. Κάναμε τη συζήτηση για τα κατόφλια και το χρονοδιάγραμμα για την ανακατάταξη. Αυτά κινούνται στη σωστή ατραπό. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετό χρόνο για τους λιανο, λιανεμπόρους, ε, ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τα νέα, τις νέες απαιτήσει των, α, της νέας ταξινόμησης και παράλληλα θα δίνουμε και τους, α, τις σωστές προφορίες στους καταναλωτές. Τρίτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι αρχές εποπτείας αγοράς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλοι ξέρουμε ότι σε διαφορετικά κράτη-μέλη αυτές οι αρχές ε, δεν έχουν αρκετά δεν είναι αρκετά καλά επανδρομένες, δεν έχουν προσωπικό και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το διευκολύνουμε, με τη χρήση μιας βάσεως δεδομένων. Να έχουμε ένα κεντρικό ε, σύστημα που το διαχειρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ εναλλακτικά είπα. Οι πληροφορίε α μείνουν στου παραγωγού και οι αγορέ, ε, εποπτείε αγορά μπορούν μέσω μια ε, διεπαφή να έρθουν σε να ρωτήσουν πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. Και έτσι όλοι οι πάντες, οι κομισιόν, οι αρχές ε, εποπτείας της αγοράς, η παραγωγή κτλ. μπορούν να έρχονται σε επαφή με αυτόν τον τρόπο. Μέσω της διεπαφής δηλαδή απευθύνονται όλοι στην βάση των δεδομένων ή στις βάσεις των δεδομένων να υπάρχει ένας κανονισμός πλαίσιο, αυτό είναι βασική φιλοσοφία, να υπάρχουν ξεκάθαρα μηνύματα ε, στους ε, καταναλωτές για να παίρνουν σωστές αποφάσεις για τις ρυθμιστικές αρχές αν θα πρέπει να ελέγχουν και τι θα πρέπει να ελέγχουν και να υπάρχει λοιπόν κάτι το πολύ ευέλικτο, μια περίοδος έτσι μετάβασης, πολύ εύκολη ε, για να περάσουμε ομαλά στο νέο σύστημα. Αυτά είναι οι βασικές προτεραιότητες της ομάδας μου. Ο κ. Ηλικιώτης από την ΚΟΕ, που είναι συντονιστή και σκιώδη εισηγητή. Και τα δύο μαζί. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχικά ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο Νοτάρο Ταμπουράνο, για την πολύ καλή δουλειά που έκανε με τι συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά και βέβαια και τη συνεχή προσπάθεια του ιδίου και όλων των σκιώδων εισηγητών για να έχουμε μια ε, καλύτερη συνεργασία όλε οι πολιτικέ ομάδε και να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ε, οι τροπολογίε που κατέθεσε η ομάδα μα, η ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, στοχεύουν στι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν στο σύστημα επισήμανση ώστε να επιτευχθεί η αύξηση τη ενεργειακή απόδοση αλλά και η ενίσχυση τη προστασία και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, εμεί όπω και άλλοι ιδέε υποστηρίζουμε πω πρέπει να διαγραφούν τα σήματα που παραπλανούν του καταναλωτέ, όπω για παράδειγμα τα συν συν συν, και να υπάρξει ένα απλούστερο ενιαίο σύστημα ανεπισήμασης από το A ως το G έτσι οι θα έχουν σαφέστερε ενδείξει για την ενεργειακή απόδοση ενό προϊόντο και θα είναι σε θέση να κάνουν συνειδητέ επιλογέ, με τις οποίες να εξοικονομούν ενέργεια αλλά και χρήματα. Η πρόταση για το σύστημα G σε συνδυασμό με την πρόταση για ανακατάταξη όλων των προϊόντων στην κλίμακα βάσει πιο αυστηρών κριτηρίων κατά την άποψή μας θα συμβάλλει καθοριστικά και στην πρόθεση της καινοτομία για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς θα ασκηθούν πιέσεις στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, οι οποίοι θα στοχεύσουν στην κατάξυση των προϊόντων τους στο επίπεδο A. Όσον αφορά το, το χρονοδιάγραμμα για την έναξη της ανακατάξη των προϊόντων στην κλίμακα, θεωρούμε πως πρέπει να αρχίσει άμεσα ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου λόγω των υφιστάμενων ελαστικών κριτηρίων το 40% των προϊόντων βρίσκεται στις τάξεις A και B της κλίμακας. Εξίσου σημαντική για την ενωτική αριστερά είναι η πρόταση για δημιουργία μιας νέας ψηφιακής βάσης δεδομένων για τα προϊόντα στην οποία όλοι οι καταναλωτές να έχουν δωρεάν πρόσβαση. Η βάση αυτή πρέπει να δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές για τα προϊόντα πέραν αυτών που αναγράφονται στην ετικέτα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και τέλο, πρέπει να παρέχει συμβουλέ ω προ τα δικαιώματα των καταναλωτών σε περίπτωση απάτη. Έτσι θα πετύχουμε να τεθεί φραγμό στην εσφοκέντρια αλλά και στην παραπλάνηση των καταναλωτών από τι μεγάλε επιχειρήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, uh, thank you very much, colleague, for your... Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Κυρία Μποναφέ, ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι μια έκθεση πλαίσιο πολύ σημαντική. Και η παρουσίαση πάνω από 700 τροπολογίες, όπως είπε ο ο Σταμπουράνο, ε, το αποδεικνύει. Δείχνει πόση σημασία δίνει το Κοινοβούλιο για αυτή την πρόταση και πόση επίγνωση υπάρχει ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τη βιομηχανία, αλλά και την αγορά τελικά. Κατά τα άλλα, είναι μια πρόταση που πρέπει να ειδωθεί μέσα σε ένα πλαίσιο με σκοπό να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση ε, βάσει της δεσμεύσης που έχει λάβει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και έναντι του έξω κόσμου και θα πρέπει να επιτρέψει, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, την ε, υιοθέτηση επιλογών με μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από τους καταναλωτές και να δοθούν και κίντρα επίσης ε, στην, καινοτομία, ε, προς την, στην βιομηχανία προς την καινοτομία με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή απόδοση χωρίς όμως γραφειοκρατία και χωρίς επιπλέον κόστος. Από την άλλη, για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα δεν μας μένει παρά να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην έρευνα, στην ποιότητα των προϊόντων που σέβονται την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όλα αυτά τα θέματα τα θίγει αυτή η πρόταση, η, πρόταση, η βάση δεδομένων. Και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θέλουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τον καταναλωτή. Τώρα θέλω να μπω πιο βαθιά σε δύο θέματα που με ενδιαφέρουν πολύ, γιατί τα θεωρώ πολύ σημαντικά ένα από τα πιο ευαίσθητα ή ίσως το πιο ευαίσθητο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγάλη προσοχή είναι το θέμα της ανακατάταξης των προϊόντων στις κλίμακες. Είμαι σκιώδης για την ομάδα μου. Η περιοδική αναθεώρηση των ετικετών πρέπει να είναι μια έξυπνη διαδικασία και θα πρέπει να έχει σαν στόχο πάνω απ' όλα να κρατήσουμε τις ενεργειακές κατηγορίες των προϊόντων ε, κατανοητές και έβλεπτες από τους καταναλωτές. Αυτό είναι το σημείο. Με βάση τη σημα... την πραγματικό των προϊόντων που είναι παρόντα στην αγορά, να καταλάβουμε τι διαφοροποίηση υπάρχουν, κυρίως ε, για τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν μεγάλη ε, ενέργεια. Κυρίως, ας πούμε, ε, οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψήξης. Επομένως, θα πρέπει να καταλάβουμε για κάθε ομάδα προϊόντων τι συμβαίνει, και να μην ε, καταλήγουν στην ίδια κατηγορία προϊόντα που έχουν ενεργειακή απόδοση πολύ διαφορετική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταλαβαίναμε την, ε, τις κλίμακες ενεργειακές, η κλίμακα θα έχει καμία σημασία και δεν θα υπήρχε καμία μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά για τον καταναλωτή. Αντίθετα, ο στόχο μα αυτό είναι. Μεγαλύτερη διαφάνεια για τον καταναλωτή. Δεύτερον, και αυτό είναι το άλλο σημείο το οποίο θέλω να αγγίξω, ε, κάτι πιο έτσι μακρόπνο, νομίζω ότι σε αυτό το κείμενο και πρέπει, πρέπει και μπορούμε ούτως ώστε να συνάδει με την δράση μας ε, στους άλλους τομείς ε, που είναι το κλίμα, η ενέργεια και το περιβάλλον. Ε, να λάβουμε υπόψη μας τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Είναι σημαντικό στην πρόταση αυτή να βάλουμε και πληροφορίες επιπλέον για την χρήση των πόρων, τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, τη δυνατότητα να επιδιορθωθούν τα προϊόντα κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλο uh, Άλλος της, αγορεύει βούλετε. Λοιπόν, η κυρία Μέρι Ντόναλη, διευθύντρια της DG Energy, ας προβεί σε κάποια σχόλια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε τον λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να πω μερικά λόγια απόψε. Ακούσαμε με τα μεγάλης προσοχή τα σχόλια του εισηγητού και των σκιωδών εισηγητών. Ευπρόσδεκτες οι προσπάθειες, οι αξιέπαινες προσπάθειες του εισηγητού να προωθήσει το θέμα. Συμμεριζόμαστε μαζί σας έναν κοινό στόχο. Με το νομοθέτημα θέλουμε να πετύχουμε ε, αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα σωστά εντοπίστηκε από τον κύριο Ρόιλ. Θέλουμε μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και από αυτή τη βάση να εξοικονομήσουμε χρήματα για τον καταναλωτή. Πρώτη προτεραιότητα που θέλουμε να πετύχει το νομοθέτημα. Ο μηχανισμός που προτείνει η νομοθεσία είναι να έχουν πληροφορίες οι καταναλωτές, βάσει των οποίων μπορούν να κάνουν την επιλογή τους. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν η ίδια επιλογή όταν θέλουν να αγοράσουν κάτι βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών. Στηρίζουμε έτσι τους καταναλωτές, που είναι βασικοί παράγοντες της αγοράς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσουμε τη σύγχυση στο νου του καταναλωτού. Αυτό σημαίνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την κυρία Ντάρλινγκ και τον κύριο Σιλικιώτη ότι θέλει αλλαγή της κατηγοριοποίησης και η ετικετοθεσία θα πρέπει να γίνει γρήγορα ούτως ώστε να μην παρατείνουμε συνδυασμό ετικετών, πολλαπλές ετικέτες που υπάρχουν στην αγορά και που δημιουργούν σύγχυση για τον καταναλωτή. Τώρα οι άλλες ταξινόμησεις και πώς θα γίνουν οι αλλαγές κατηγοριών, αυτό είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, μετά από συζητήσεις σχετικά με τη βάση δεδομένων. Πραγματικά πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ποια είναι η λογική μας όταν προτείναμε τη βάση δεδομένων. Θέλαμε καλύτερη ρύθμιση. Αυτή την προσέγγιση ακολουθήσαμε. Είδαμε το διοικητικό κόστος και το άχθος για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο και σε αυτόν και σε άλλους τομείς. Και είδαμε και στους τίτλους εφημερίδων άλλους τομείς για δραστηριότητε η έλλειψη αυτών. Θέλαμε να υποφεληθούμε από τις νέες τεχνολογίες για να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τα κράτη-μέλη όσον αφορά επαλήθευση συμμόρφωσης κλπ. Και δεύτερον, να γίνει διαφανέστερη η πληροφορία, να διατίθεται στους καταναλωτές για τα προϊόντα. Χαιρόμαθα ιδιαίτερος να ακολουθήσουμε την πρόταση του κ. Πέταλε όσον αφορά τι χώρε που θα έχουν τυποποιημένη σελίδα που θα διατίθεται και θα είναι προσβάσιμη εύκολη. Αν είναι ρεαλιστικό θα το κάνουμε. Εάν είναι η πρακτική λύση α την ακολουθήσουμε. Αν όχι θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε μια ενιαία θηρίδα αν θέλετε για ενημέρωση των καταναλωτών στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου στον οποίο ζούμε. Και στο κείμενο και στην ανάλυση που προηγήθηκε του κειμένου εκτιμήσαμε το ετήσιο κόστος αυτού και για την κλίμακα της ευρωπαϊκής αγοράς το κόστος είναι αρκετά λογικό σχετικά με τις γλώσσες για το έγγραφο Πιστεύω ότι η δεθεσιμότητα της τεχνολογίας θα μας επιτρέψει σημαντικά σε αυτό τον τομέα. Έχουμε αυτόματα συστήματα μεταφράσεως και έτσι ο καταναλωτής θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες ανεξάρτητα από τη γλώσσα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Α, προχωρά το θέμα πάρα πολύ καλά, χάρη στη σκληρή δουλειά του, του εισηγητού και των άλλων μελών. Πιστεύω ότι έχουμε ενόψει πολύ ρεαλιστικές τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα μπορέσουμε να το προωθήσουμε και να ολοκληρωθούν συντομότατα οι εργασίες μας. Είναι κάτι που θέλουν να έχουν γρήγορα στα χέρια τους ε, οι καταναλωτές τη Ευρώπη και να το λάβουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γενική Διευθύντρια. Ο εισηγητή μας, ο συνάδελφός μας, ο κύριος Ταμπουράνο. Κύριε Ταμπουράνο, έχετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σκέψεις που εξέφρασαν. Θα είμαι πολύ σύντομος θα ήθελα να τονίσω κάτι που τονίζω. Η εποπτική αρχή, η εποπτικός φορέας της αγοράς. Λοιπόν, δεν υπάρχει αντιστοιχία στον αφορά των έλεγχο της αγοράς όταν κάτι μελη Κάποια κάτι έχουν περισσότερους πόρους, άλλα κάτι πολύ, λίγες, ε, πολύ λίγους πόρους και πιστεύω ότι ο καλύτερος δρόμος για να βελτιώσουμε τη διαδικασία της εποπτείας του αγοράς είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών, πραγματικά αυτή να αποφύγουμε κάθε αγορά της αγοράς να μην γνωρίζει τι κάνει η άλλη και ο τρόπος με λιγότερους πόρους λόγω συνεργασίας σίγουρα θα βελτιώσουμε την αποδοτικότητα τη γενική σε επίπεδο 28 κρατών μελών. Όσον αφορά την database, τη βάση δεδομένων, ας πούμε ότι αυτή η Επιτροπή της Βιομηχανίας ασχολείται με θέματα βιομηχανίας και ενέργειας και για να ξαναπροθίσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειαζόμαστε κάποιο βαθμό ανταγωνιστικότητας και δεν μπορούμε να μένουμε πίσω σε σύγκριση με άλλους παγκόσμιους φορείς όπως είναι η Αυστραλία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Κίνα ακόμα που ήδη έχουν βάση δεδομένων προϊόντων. Εμείς είμαστε μια μεγάλη δύναμη σε πλανητικό επίπεδο και πιστεύω δεν μπορούμε να υπολοιπόμεθα αυτόν. Αυτή η βάση δεδομένων θα μπορεί να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα το ιδιαίτερο της υπήρου μας, που είναι η πολυγλωσία. Έχουμε τις τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και το να, να περάσουμε από χάρτινες οδηγίες σε ψηφιακές οδηγίες νομίζω είναι σωστός δρόμος για να το πετύχουμε αυτό. Τώρα, ως... Δηλαδή, να περάσουμε από χάρτινες οδηγίες σε ψηφιακές οδηγίες θα βοηθήσει να μειωθεί και το βάρος ε, της βιομηχανίας. Πράγματι, μια πρώτη αλλαγή κλίμακας και η δρομολόγηση της βάσης δεδομένων ίσως να είναι μεγάλο βάρος, αλλά αυτός ο μεγάλος κόπος, αυτή η μεγάλη κατανάλωση δυνάμεων και ανθρωπίνων πόρων θα μπορούσε να αντισταθμιστεί ακολούθως ε, για να γίνει πιο ρευστή όλη η διαδικασία και σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος Βοναφέ, να βάλουμε υπόψη ότι η ψηφιοποίηση είναι μίες, μία από τις διαδρομές που μπορεί να μας οδηγήσει πιο εύκολα προς την κυκλική οικονομία. Δηλαδή να γίνουν άειλες οι πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για την έκθεσή σας, για τη σκληρή δουλειά σας Όσον αφορά τις τροπολογίες, συμβιβαστικές τροπολογίες, να σας πω ότι η ψηφοφορία στην Ήτρε προβλέπεται 24 Μαΐου, ενεστώτος έτους βέβαια, σε έξι εβδομάδες λίγο πολύ. Στην Ολομέλεια θα δούμε πότε θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Τελειώσαμε το σημείο 11. Να υπογραμμίσω ότι είμαστε λίγο πιο γρήγοροι από ό,τι είχαμε προβλέψει. Κάποιοι από τους συναδέλφους μας είχαν προβλήματα να βρουν εισιτήρια για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και έπρεπε να αποχωρήσουν ακόμα και να φύγουν το πρωί. Οπότε στις 10 στην ψηφοφορία είχαμε λιγότερους από 67 συναδέλφους που ψήφισαν. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία μας. Πάντα είχαμε 75, 72, αυτή τη φορά είχαμε λιγότερους από 67 παρόντες. Γι' αυτό προχωρούμε κάπως πιο γρήγορα και ίσως αυτό να βολεύει και άλλους συναδέλφους, διότι κάποιοι από εμά πρέπει να φύγουμε στις 5 ή στις 5 και μισή, άρα χρειάζεται να είμαστε και στα αεροδρόμια στις Βρυξέλλες τουλάχιστον μία μισή με δύο ώρες νωρίτερα πριν την αναχώρηση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις εργασίες μας. Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, σημείο 12. Να σας πω ότι στην έκθεση, την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας αυτή βασίζεται σε ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας. Να υπενθυμίσω σε όλους σας το σχέδιο εκθέσεως υπευλήθη στις 22 Φεβρουαρίου και να σας πω επίσης ότι υποβάλαμε 448 τροπολογίες. Η κυρία Τερέζα Γκρίφιν είναι η συγγητριά μας. Είμαι ήρεμο για την κατάσταση, διότι η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ είναι εδώ μαζί μα και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αντικαθιστώ πολλού συναδέλφου σήμερα το απόγευμα λόγω των προβλημάτων με τα ταξίδια. Η Τερέζα δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί, ζητάει συγγνώμη. Θα διαβάσω λοιπόν μία δήλωσή της. Αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα μας, σοσιαλιστές και δημοκράτες και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Στόχος της να τονίσει το ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης. Εν γέννη πιστεύουμε ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να έχει τα συμφέροντα των πολιτών στο κέντρο της και σαν γενική αρχή η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να καταλήξει σε πιο αποκεντρωμένο δημοκρατικό ενεργειακό σύστημα που είναι υποφελές για όλη την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα για να πετύχουμε πραγματικά ανταγωνιστική αγορά λιανικής που θα είναι φιλική του καταναλωτή. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια για του λογαριασμού και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι πιο εύκολο να συγκρίνουμε συμβάσει και προσφορέ για όλου του καταναλωτέ που προφανέ αυτό συμπεριλαμβάνει και εκείνους που δεν γνωρίζουν καλά τα τέλη, δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ. Δεν είναι καλά πληροφορημένοι. Ζητά οι προμηθευτές, ζητά έκθεση να δίνουν οι προμηθευτές τους καταναλωτές για τις καλές προσφορές και να ενημερώνονται και για τις τιμές των ανταγωνιστών. Θα πρέπει να απαγορευτεί η αθέμητη εμπορική πρακτική, διότι βλέπουμε αύξηση καταγγελιών όσον αφορά πώληση από πόρτα σε πόρτα και ε, παράξενους τρόπους ε, marketing στα κάτι μέλη. Λοιπόν, στο πλαίσιο τη ενεργειακή μετάφαση θα πρέπει να βοηθήσουμε του καταναλωτέ να ε, εστερνιστούν την αλλαγή, να έρθουν τα εμπόδια, ώστε να μπορέσουν να παράξουν τη δική του ενέργεια και να έχουν, πετύχουν ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να προωθήσουμε και την ανάπτυξη ανταπόκριση στη ζήτηση, εξασφαλίζοντα ότι η ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών δεν θα αφήσει του πλέον ευάλωτου ή λιγότερο ε, εξοικειωμένου καταναλωτέ πίσω. Για την καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια, ε, που είναι κάτι που θέλει να πετύχει η Τερέζα, πιστεύουμε ότι πέρα από τι κοινωνικέ πολιτικέ ε, και με μέτρα ενεργειακή απόδοση για του ευάλωτου ε, πολίτε είναι κάτι σημαντικό. Και η ανανέωση των κτηρίων είναι ένα καρπό που είναι εύκολο να δρέψουμε. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει σχέδιο δράση για την ενεργειακή φτώχεια και θα πρέπει να έχει σε στόχο την ενεργειακή απόδοση βάσει υποχρεώσεων για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενέργειας. 4.048 ε, ε, τροπολογίες υπευλήθησαν και διατρέχουμε όλες τις τροπολογίες μαζί με τους σκιώδεις προσπαθώντας να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες. Η Τερέζα θέλει να ευχαριστήσει όλους τους σκιώδεις ηγητές για την καλή του συνεργασία μέχρι τώρα. Θα λάβει υπόψη και αυτή και η ομάδα της όλα τα σχόλια τα οποία θα ακουστούν σήμερα και σαν ομάδα προσβλέπουμε σε συνεργασία με όλους ώστε να ολοκληρωθούν οι συμβαστικέ λύσει και να αναπτύξουμε μια ισχυρή στεναρή έκθεση που θα προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανταποκριθούμε στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το ΕΛΚ. Ο Σον Κέλλη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την συνάδελφο που ανέπτυξε τις απόψεις της ε, κυρίας Γκρίφιν την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει κάνει και για την διάθεση συνεργασίας. Νομίζω πως είμαστε κοντά σε μια αποδεκτή θέση για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση της Επιτροπής μας. Νομίζω πως όλοι οι σκιώδεις ε, συμφωνούν στο βασικό στόχο δηλαδή να έχουμε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να εμπλακούν στην αγορά ενέργειας. Νομίζω λοιπόν πως πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχουν ακουστεί ε, ενδιαφέρουσες ιδέες. Το βασικό σημείο εδώ πέρα είναι πως ε, θα γίνει μια νέα συμφωνία με τους καταναλωτές για μια αγορά που θα λειτουργεί σωστά. Η διαφάνεια, οι συγκρίσιμες τιμές και οι πιο ενημερωμένοι καταναλωτές ε, αποτελέσουν θετικά σημεία. Θα δούμε αλλαγές στα ενεργειακά συστήματα, θα έχουμε αποκεντρωμένη παραγωγή. Τώρα οι καταναλωτές ε, θα επενδύσουν σε μικροεγκαταστάσεις παραγωγής για να αρχίσουν να παράγουν τη δική τους ενέργεια είναι μια θετική εξέλιξη που θα μειώσει τις εκπομπές, θα αυξήσει τις ανανεώσιμες και θα πετύχουμε τους στόχους. Ειδικά στη δική μου την περιφέρεια υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής των πολιτών και παραγωγής ε, ανανεώσιμης ενέργειας ε, και νομίζω πως έτσι θα αυξηθεί η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και Βεβαίω θα επηρεαστούν και οι ανεμογεννήτριε που αυτή τη στιγμή περνάνε μια δύσκολη φάση στη χώρα μου. Το το οποίο όμως τονίζουμε είναι όλο και πιο αποκεντρωμένη παραγωγή. Έχει σημασία η σταθερότητα του δικτύου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας αποτρέπει από την ε, παραγωγή μικρής κλίμακας. Ε, όμως οι ε, ανατόμες τεχνολογίες θα χρειαστούν για να πετύχουμε αυτή την ευελιξία. Νομίζω πως αυτό θα είναι βασικό κομμάτι της έκθεσης Λάγκεν για το σχεδιασμό της αγοράς. Η ενδυνάμωση των καταναλωτών είναι σημαντικό κομμάτι όλων αυτών. Θεωρώ ότι έτσι θα μπορέσει να ζητήσει τα καλύτερα συμβόλαια ο καταναλωτής Θα πρέπει λοιπόν ο καταναλωτής να είναι πιο ενεργός και βεβαίως η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τιμών θα μπορέσουν να οδηγήσουν τους ενημερωμένους καταναλωτές στην καινοτομία. Είναι μια κατάσταση από την οποία αποφελούνται όλοι. Και έτσι θα υπάρχει δυνατότητα στο κρατών μέλο, στα κράτη-μέλη να ενημερώνονται οι καταναλωτέ για φόρους και τέλη που ενσωματώνονται στην τιμή τη ενέργεια και έτσι θα υπάρχουν ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης ε, των τιμών ε, που μπορεί να είναι και ε, μέρος κάποιων άλλων φορέων όπως τα Υπουργεία ενέργεια. Αν θέλετε μπορώ να σταματήσω να ξεπεράσω το χρόνο. Δεν σταματήσα κανέναν, λέει ο πρόεδρος. Και ελπίζω να μην ε, ξεκινήσουμε τώρα με δεκάλεπτες ομιλίες. Έχετε, έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ λοιπόν. Καλώς ορίζω το ότι η συγγήτρια ζητάει να κινητοποιηθεί η ομάδα εργασίας έτσι ώστε οι τιμές λιανικής να ανταποκρίνονται κάπως στις ε, τιμές χονδρικής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αντικατοπτρίζουν την προσφορά και την ε, ζήτηση. Η τεχνολογία της πληροφορικής είπα, θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή. Συμπερασματικά θεωρώ πως τώρα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε σε μια ανταγωνιστική και διάφανη αγορά η οποία θα μειώσει το κόστος της ενέργειας και έτσι θα αυξηθούν οι δαπάνες των οικοκυριών και άρα θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Οι χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας σημαίνει ότι θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες κατανάλωσης ε, οι πολίτες και άρα θα ωφεληθούν και οι επιχειρήσεις. ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι τους ε, εισηγητές ε, και αναμένω την συνεργασία μας σε επόμενες εβδομάδες για τους καταναλωτές και πολίτες μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η κυρία Αγγέλ Μίλλερ. Αλλά ο Φίλιπ Τεμπάκερ είναι έτοιμος για τα πάντα, για να αντεκαταστήσει τους πάντες παρότι κρύβεται πίσω από την, το προσωπείο της Αγγέλικα. Είναι μεγάλη η Αγγέλικα. Μιλάω εξ ονοματός της. Είναι... Ναι. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους και εισηγητές για την καλή συνεργασία. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ε, προχωράει απρόσκοπτα για μια ισορροπημένη έκθεση και θέλει να τονίσει ότι οι καταναλωτέ θα πρέπει να είναι στο κέντρο τη ενεργειακή μετάβαση. Οι τροπολογίε τη Αντζέλικα και τη ομάδα μα τονίζουν τη σημασία τη ενίσχυση των καταναλωτών, τη ενδυνάμωση των καταναλωτών να παίρνουν ε, καλύτερε επιλογές μέσω τη καλύτερη ε, ενημέρωση, τη μεγαλύτερη προστασία του, αλλά θέλει επίση να έχουν τη δυνατότητα να είναι ενεργοί συμμέτοχοι στην ε, αγορά, η παραγωγή, οι ενδιαφερόμενοι όλοι μαζί με τους καταναλωτές, ε, τα μηχανισμοί χρηματοδότησης, ε, μπορούν όλοι οι φορείς μαζί να συνεισφέρουν καλύτερα και να βοηθήσουν σε αυτή τη μετάβαση. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ενεργειακό σύστημα από πίσω, το οποίο θα πρέπει πάνω απ' όλα να λειτουργεί. Ούτως δεύτερον, για να έχουμε πιο αποκεντρωμένη και ευέλικτη αγορά, θα πρέπει να βελτιωθεί η συμμετοχή των ε, τοπικών αρχών, των πόλεων. Είναι ο κρίκο πιο κοντά στου πολίτε από εκεί ξεκινάει η οντομία και η Κομισιόν υποστηρίζει τη συνεργασία του, των δημάρχων μέσω του συμφώνου των δημάρχων και αυτό θα είναι βασικό εργαλείο για να πετύχουμε αυτή τη συνεργασία. Ένα άλλο σημείο για μα είναι οι έξυπνε τεχνολογίε για να εμπλέξουμε ενεργά του καταναλωτέ και να του βοηθήσουμε να μειώσουν την κατανάλωση και το κόστο κατανάλωση, ούτω ώστε να υπάρχει ένα σύστημα πιο ενσωματωμένο ζήτηση και παροχής ε, και να λάβουμε υπόψη μας και τις επενδύσεις που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ε, θα έχουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε, να έχουμε έξυπνες, έξυπνους μετρητές, κινητές εφαρμογές κτλ. ή εφαρμογές στα κινητά. Μέχρι στιγμής 16 κρατημέλη έχουν τους έξυπνους μετρητές, πολλά κρατημέλη καθυστερούν. κάνουν ακόμα μία ανάλυση κόστους-οφέλους ενώ τα ωφέλη είναι σαφώς ε, εδώ μπροστά μας. Τι περιμένουμε λοιπόν. Ε, επίσης οι έξυπνες συσκευέ θα παίξουν το ρόλο τους να υπάρχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα ούτως ώστε οι καταναλωτές να ε, δρέψουν πλήρως τα ωφέλη. Ε, Κύριος Γιαβόρ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαραγάλ κανονικά θα ήταν ο εισηγητής, αλλά ζητά συγγνώμη λόγω των προβλημάτων με τα ταξίδια. Δεν μπορεί να είναι εδώ παρόν το απόγευμα. Καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Γκρίφιν για την καλή συνεργασία. Ελπίζουμε ότι η συνέχιση αυτής της συζήτησης θα οδηγήσει σε μια κοινώς αποδεκτή λύση, ένα καλό έγγραφο η Κομισιόν λέει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι στο κέντρο της Ενεργειακής Ένωσης. Ε, και έχουμε και την ανακοίνωση για τη νέα συμφωνία για, για την ενεργειακή κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε ένα κεντρικό σύστημα και θέλουμε να περάσουμε σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα, ε, να δώσουμε εξουσία στους ε, καταναλωτές, να περάσουμε από το από την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, χάρη στη φοβερή μείωση του κόστου των ανανεώσιμων. Έχουμε διαδικασίες αδειοδότησης. Ε, δεν πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις για τις υπερβάσεις. Ε, θα πρέπει τα τιμολόγια να βασίζονται ε, στο δυναμικό και όχι, ή μάλλον βασίζονται στο δυναμικό και όχι στην κατανάλωση και αυτό αποθαρρύνει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό δείχνει πω σημαντικό οι πολίτε να είναι στο κέντρο τη Ενεργειακή Ένωση και να μην μείνει αυτό ένα κενό ε, σλόγγαν. Γι' αυτό οι πράσινοι θέλουν μια απλούστευση τη διαδικασία συμμετοχή των καταναλωτών και νοικοκυριών μέσω τη μελλοντική νομοθεσία για την ενέργεια και να ληφθεί υπόψη η επίπτωση που θα έχει σε αυτού ε, από την Ενεργειακή Ένωση. Η πρόσβαση σε αξιόπιστη και διαφάνεια, ε, διαφανή πληροφορία σε ό,τι αφορά τις, ε, ε τα τιμολόγια, ε, σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις κτλ. Ούτως ώστε να κάνουν ε, εγνωσμένες επιλογές οι καταναλωτές. Τρίτον, μεγάλο μέλημα για μας είναι η δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου για την ενέργεια. θέλουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πραγματικά θα ενισχύει τους ε, πολίτες και τους κάνει ενεργούς μετόχους στην αγορά ως ε, ενδιαφερομένους αλλά και ως επενδυτές. Να έχουν το δικαίωμα να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια σε δίκαιες τιμές. Να, ε, επίσης να αρθούν τα διοικητικά φράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ούτως ώστε να είναι πιο αξιόπιστο το περιβάλλον για την αυτοκατανάλωση ενέργειας, αν θέλετε να περάσουμε στη νέα ενεργειακή φάση ε, με επιτυχία. Ε, για να το κάνετε αυτό όμως πρέπει να δώσετε εξουσία στους ίδιους πολίτες. Ευχαριστώ συναδελφοί. Κυρία Κάλλας είναι υπεύθυνη. Ο κ. Μπενίτο Ζιλουάγκα, σκιώδη τη Γκουε. Η επόμενη είναι η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε σε μια πρώτη φάση. Έδειξε δύο πράγματα που μας φαίνονται πολύ σημαντικά. Σε μια πρώτη φάση, τη θέληση να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στους οικιακού χρήστες ενέργειας σε αυτή την έκθεση, ε, γιατί αυτοί χρειάζονται πάνω απ' όλα τη δική μας δράση, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ε, εμπορικές καταχρήσεις και από την άλλη θα πρέπει να εκδημοκρατικοποιηθεί το ενεργειακό σύστημα για να συμμετάσχουν πιο απρόσκοπτα οι καταναλωτές και η παραγωγή. Για το τελευταίο κομμάτι όμως αυτό, δυστυχώς η έκθεση παρουσιάζει ελλείψεις και κενά. Γιατί ε, εδώ άφησε το αποτύπωμά της η δεξιά, δυστυχώς. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό το δεύτερο κομμάτι και πρέπει να πάμε πιο τα εκεί. Όταν μιλάμε για ενεργειακή μετάβαση, δεν μιλάμε μόνο για, λιγότερο, για λιγότερη κατανάλωση και περισσότερου ηλιακού θερμοσυσσωρευτέ. Και αυτά σημαντικά. Η ενεργειακή μετάβαση σημαίνει να περάσουμε σε ένα μοντέλο πιο ισοσκελισμένο, ας πούμε. Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, πηγών ενέργειας. Μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για την ενεργειακή φτώχεια εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά, αλλά δεν, αν δεν δούμε τα ιδιωτικά συμφέροντα σε αυτό το κύκλο της ενέργειας, δεν έχει νόημα. Ε, έχουμε, όταν υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω νέων ε, καινοτόμων μοντέλων, όπως λένε κάποιες τροπολογίες, σημαίνει ότι ανοίγουμε την, πόλα, την πόρτα στο ιδιωτικό κεφάλαιο, που εξορισμού ψάχνει το κέρδο και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να προωθήσει τους κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους. Για μας λοιπόν ε, παραμένει ενισχύει η πρόταση, η πρόταση ότι οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να μπαίνουν στον υπολογισμό του ελλείμματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα κράτη-μέλη και για τη στρατηγική που θα αναπτύξουν. Τις τελευταίες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χρησιμοποιηθεί αυτή η φόρμουλα για, τους, για τις δαπάνες και το, το πρότεινε ε, κυρίως για ορισμένους τομείς, κυρίως για το στρατιωτικό. Γιατί να μην το προτείνει γενικά αυτό όμως. Ευχαριστώ συνάδελφε κυρία Κάλλας που ετοιμάζει γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΕΜΚΟ στο ίδιο θέμα για αυτή την προσφορά για τους καταναλωτές ενέργειας. Ναι, ήμουν εισηγήτρια στην ΕΜΚΟ για το ίδιο θέμα. Η γνωμοδότηση ήδη θετήθηκε. Μόνο δύο ψήφοι κατά, καμία αποχή είναι σύντομη. Η κυρία Γκρίφιν ελπίζω να λάβει υπόψη της τους σχετικούς συμβιβασμού σχόλια. Στην έκθεσή της, η κυρία Γκρίφιν συνδέει άμεσα το να δώσουν δυνατότητε στους καταναλωτές και έτσι να γίνουν συνειδητοί καταναλωτές. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό όλοι οι καταναλωτές. Δεν θέλουν την ίδια εμπλοκή στις προσπάθειε εφοδιασμού ενέργεια θα μπορούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια σε διαφορετικό επίπεδο. Πρέπει να γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Για να δώσουν περισσότερε δυνατότητε στου καταναλωτέ, χρειάζονται πληροφορίε για να αποφασίσουν. Σε πραγματικό χρόνο, για την κατανάλωση μέσω εφιών εργαλείων πληροφορική, σωστέ πληροφορίε για του λογαριασμού κατανάλωση ενέργεια. Δεν είναι σωστό αυτές οι πληροφορίες να λαμβάνονται μία φορά το χρόνο, κάτι που ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη. Στην Εστονία κάθε μήνα. Να δίνονται συχνά οι λογαριασμοί, να καταλαβαίνει ο κόσμος και στο λογαριασμό να φαίνονται ακριβώς ε, τι χρεώνονται. Πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή κόστους μεταξύ των καταναλωτών των ε, ε, εκείνων που πληρώνουν και για το δίκτυο και των πιο επαγγελματιών, των που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Χρειάζεται ισορροπία στο δίκτυο. Και οι δικαιώματα και οι υποχρεώσεις είναι ισορροπημένα. Για τα δεδομένα. Η συμβαστική 36 της παραγράφου 20. Ερώτηση για τη συγκήτρια. Προσωπικά στοιχεία, τι εννοούμε. Όνομα και διεύθυνση ή στοιχεία που αφορούν την προσωπική χρήση ενέργειας. Στην τροπολογία μου ξεκαθαρίζω ότι η χρήση των δεδομένων πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο προστασία των δικαιωμάτων. Δικαίωμα πόση συνένεση, παραδείγματο χάρη. Όταν μιλάμε το δικαίωμα διαγραφή στοιχείων, πρέπει να καταλάβουμε το πλαίσιο. όπου εκείνοι που κάνουν χρηση εντάσετε στο στην φορείς διανομής πρέπει να εντασσεται στο πλαισιο προστασια των δικαιωματων δικαιωμα ποση συνενεση παραδειγματο χαρη οταν μιλαμε το δικαιωμα διαγραφη στοιχειων πρεπει να καταλαβουμε το πλαισιο οπου εκεινοι που κανουν οι φορει διανομη πρεπει να εχουν τα σωστά στοιχεία για να διαχειρίζονται το δίκτυο. Όταν μπορεί κανείς να αποσύρει τα στοιχεία, τότε καταρρεί το σύστημα. Το δικαίωμα να εισμονηθεί κανείς στο δίκτυο, στο διαδίκτυο δεν είναι το ίδιο όσο, όπως η διαγραφή στοιχείων για τη χρήση του δικτύου. Ευχαριστώ. πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τμήματάρχης ε, κυρία Αννα Κολούτση από τη Γενική Διεύθυνση Ενεργείας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επιτά μέλη της Επιτροπής ενδυνάμωση των ε, καταναλωτών είναι βασικό κομμάτι της νέας συμφωνίας με τους καταναλωτές. Βλέπουμε πως οι καταναλωτές θέλουν εμπιστοσύνη, επιλογή, αλλά και απλότητα και προστασία από την αγορά. Τα ενεργειακά συστήματα από την άλλη χρειάζονται περισσότερη ευελιξία, ανταγωνισμό, αποτελεσματικότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν το μέλλον για τους στόχους μας για το 2030. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια φιλόδοξη απάντηση και η σημερινή συζήτηση νομίζω δείχνει πως υπάρχει φιλοδοξία και χαίρομαι για αυτή τη σύγκληση. δυναμική τιμολόγηση, εύκολη αλλαγή παρόχου, τοπική δράση, ανταπόκριση στη ζήτηση, αλλά και περιορισμός της ενεργειακής φτώχειας. Είναι νομίζω αυτά τα οποία υπάρχουν στην αγορά, αλλά και στην, στο κέντρο της ανακοίνωσής μας. Θεωρώ πως πρέπει να μην χάνουμε το στόχο, να παραμένουμε προσιλωμένοι στα ζητήματα των καταναλωτών, να έχουμε αποτελεσματική δράση η οποία θα βάλει τους καταναλωτές στο κέντρο της ενεργειακής μας πολιτικής. Γι' αυτό η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές εστιάζει κυρίως σε δύο ζητήματα. Την ενδυνάμωση των καταναλωτών και βεβαίως τα ζητήματα του δικτύου διανομής για να υπάρχει αυτή η απαραίτητη ευελιξία για να γίνει η μετάβαση προς ένα σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο στις ανανεώσιμες. Γι' αυτό θεωρώ πως η έκθεση και οι πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν σωστά επισημαίνουν τις ελλείψεις που υπάρχουν στους ε, τομείς αυτούς και που κάνουν το σύστημα να μην έχει ανταγωνιστικότητα και να είναι δύσκολη η αλλαγή. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις και χάρηκα με τα περισσότερα σχόλια και την σημερινή συζήτηση και αναμένω βεβαίως ε, τις επόμενες ε, συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και την τελική έκθεση που είναι ήδη πολύ ενθαρρυντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. όλα τα σχόλια σας ε, και οι παρατηρήσεις σας βεβαίως θα διαβιβαστούν στην εισηγήτρια, την κυρία Γκρίφιν. Ψηφοφορία την 21η Απριλίου. Και ένα μήνα μετά στην Ολομέλεια η ψηφοφορία πιθανότατα. Περνάμε στο επόμενο θέμα, ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και κατάργηση της οδηγίας 2008 κάθετος 92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική διαδικασία για την βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος για τον βιομηχανικό καταναλωτή. Η κυρία Κάπελ είναι η συγγήτρια. Και ο κύριος Γκέρολφ Άνεμανς θα μας παρουσιάσει την έκθεση της κυρίας Κάπελ. Ευχαριστώ, είναι ευχαρίστησή μου να ευχαριστώ την κυρία Κάπελ. Θα σας διαβάσω τη δήλωση. Ευχαριστεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την συνεργασία και αναμένει να συνεχιστεί σε αυτή τη βάση συνεργασία μας ε, για να έχουμε στατιστικά τα οποία θα είναι συγκρίσιμα και ακριβή, καθώς αυτό είναι το θεμέλιο λογικής χάραξης πολιτικής. συλλογή δεδομένων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ε, για τους τελικούς ε, καταναλωτές, για τα νοικοκυριά, μέχρι τώρα ήταν σε θελοντική βάση, αλλά με βάση με 100% ποσοστό ανταπόκρισης και τώρα σκεφτόμαστε να περάσουμε ε, στο να γίνει το σύστημα υποχρεωτικό για να μην επιδεινωθεί δε η κατάσταση και να έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα υψηλής ε, ποιότητας και θα συνεχίσουν τα δεδομένα να συλλέγονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Στόχο λοιπόν η έκθεση έχει να ξεκαθαρίσει τους ε, στόχους, ε, να υπάρξει μια διευκόλυνση των αρχών που συλλέγουν ε, και μεταδίδουν τα δεδομένα και να μην υπάρχουν παρεξήγησεις. Συνεπώς, έχουμε ένα στοιχείο που περιλαμβάνει κάποια υποστοιχεία που παραλήφθηκαν, όπως η ειδικοί φόρη κατανάλωσης. Επίσης, ο όρος ε, της χρέωσης, ε, γιατί μεταβιβάζονται αυτή τη στιγμή χρεώσεις από το δίκτυο στην ενέργεια και αντιστρόφως, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Προτείνουμε λοιπόν αλλαγές στην ανάλυση για να αντικατοπτρίζει την δομή των τιμών. Αυτά τα δύο τελευταία σημεία είναι δύσκολο να γίνουν καθώς διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το ίδιο στοιχείο της τιμής αλλού θεωρείται τέλος χρέος ή ειδικό φόρος ε, ή οτιδήποτε άλλο αναλόγως στη χώρα. Οπότε εδώ πέρα χρησιμοποιούμε μια διατύπωση η οποία ίσως δεν ισχύει για όλες τις χώρες. Ε, επιπλέον, άλλα σημεία που αναφέρουμε στην έκθεση είναι τα εξής. Η πρόταση της Κομισιόν δεν καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των τιμών, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνουν οι πάροχοι. Πρέπει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, ή τα κράτη να κάνουν αυτή την ανάλυση και να έχουν μια μεθοδολογία και να δίνουν βεβαίω και τις απαραίτητες πληροφορίες. Και βεβαίως όλα αυτά να επαληθευτούν από την Eurostat για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Δεύτερον, είναι υποχρεωτικό να δίνουν αναφορά οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές και άρα θα είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων δεδομένων των καταναλωτών και των παρόχων. Γι' αυτό οι τιμές δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται εκτός αν υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός καταναλωτών. Αυτό είναι μια πρόταση που υπήρχε και στην προηγούμενη οδηγία με το οργανισμό 223 του 2009 που ήδη προβλέπει ότι θα συλλέγονται στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, επαγγελματικής ανεξαρτησίας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας, πώς να στατεύοντας πάντα την εμπιστευτικότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εάν μια συγκεκριμένη τέτοια πρόταση θα μείωνε την αποτελεσματικότητα του κανονισμού 223. Τέλος, ε, τα στοιχεία των χρεώσεων μπορούν να αφορούν μόνο το σύνολο των καταναλωτών, ε, νοικοκυριών και μη και όχι μόνο μερικούς μήνες. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατον ε, όταν υπάρχει μια αποδεσμευμένη αγορά ηλεκτρισμού, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία των διαχειριστών του δικτύου. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες αν η χρέωση με να κλιμάκιο κατανάλωσης. Ε, καταλήγοντας λοιπόν, η κυρία Κάπελ σας ευχαριστεί πάρα πολύ και για τις προτάσεις και για την πρώτη συνεδρία των συντονιστών θα ετοιμάσει μια σειρά συμβαστικών προτάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κριστιανής Κάρινς, ο εισηγητής του ΕΛΚ. Αλλά ο συνάδελφος Μπένστον θα μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του συντονιστού, Κριστιάνης Κάρινς. Έχω την εξής δήλωση του ΕΛΚ. Για να ληφθούν σωστές αποφάσεις, χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα, συγκρίσιμα, επίκαιρα, επικαιροποιημένα. Δημιουργούμε την Ενεργειακή Ένωση και τα στατιστικά στοιχεία είναι όλο και πιο σημαντικά. Έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τη λειτουργία εσωτερική αγορά ενέργεια σκοπός του κανονισμού. Κοινό πλαίσιο. Η ανάπτυξη, παραγωγή, δημιουργή, ε, παραγωγή και σύγκριση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια και τις τιμές αυτών για νοικοκυριά και πελάτες εκτός νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας επίκαιρα εναρμονισμένα στοιχεία για τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνται στους πολίτες χρειάζεται, χρειάζονται για να παρακολουθούμε το πώς λειτουργούν οι ενεργικές αγορές των κρατών μελών. Τα στοιχεία για τους βιομηχανικούς πελάτες συλλέγονται σύμφωνα με, με οδηγία σχετική. Όμως τα στοιχεία για τα νοικοκυριά συλλέγονται βάσει εθελοντικών συμφωνιών. Ο κανονισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου βελτιώνει το παρόν πλαίσιο. Στόχος η εναρμόνιση του πλαισίου εισάγοντας νομική πράξη που καλύπτει συλλογή στοιχείων για νοικοκυριά και τελικούς καταναλωτές που δεν είναι, δεν ανήκουν στην κατηγορία των νοικοκυριών. Δύο πράγματα να πω. Πρώτον, είναι σημαντικό η παρούσα μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει για να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Δεύτερον, η συλλογή στοιχείων θα γίνει από εκείνους που θα δίνουν τις απαντήσεις, τους ίδιους τους πελάτες. Να μην αυξηθεί το άχθος. Ζητούμε τις πληροφορίες που ήδη διαθέτουν οι συμμετέχοντες στην αγορά και έτσι δεν δημιουργούμε αύξηση της γραφειοκρατίας. Δύσκολο να γνωρίζει να μην γνωρίζει η εταιρεία τι χρεώνει στους πελάτες και οι πελάτες να μην ξέρουν τι πληρώνουν. Αυτό είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προβλέπω συνεργασία για το θέμα με τον εισηγητή και τους σκιώδες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφε. Σκιώδης του ECR. Ανλίν Βανποσιούτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορώ να πω πως είμαι ικανοποιημένοι με την πρώτη πρόταση της εισηγήτριας. ειδικά όσον αφορά την καλύτερη ρύθμιση αλλά και τα ζητήματα των διοικητικών το περιορισμών του διοικητικού βάρους όσον αφορά τώρα τις πράξεις ε, κατεξιοδότηση πρέπει να το δούμε με την εισηγητρία γενικά Είμαι πεπισμένη ότι όντως χρειάζεται να έχουμε καλύτερα δεδομένα για τις τιμές της ε, ενέργειας ε, και για να ασκήσουμε μια πολιτική ευρωπαϊκή τα χρειαζόμαστε. Βλέπουμε παραδείγματο χάρη ότι η τιμή τη ενέργεια ε, κατά 50% και παραπάνω είναι φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι κατανάλωση κτλ. Οπότε θα πρέπει να δούμε και να μπορούμε να βλέπουμε ποιε είναι οι τάσει και να γίνονται ε, συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ε, η φορολογία βεβαίως είναι αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών. Και ε, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια εναρμόνιση των φόρων. Είμαι λοιπόν πεπισμένοι ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια ισορροπία με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάβολ για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω ως και ο Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Κάπελ για το σχέδιο κειμένου. Γενικά έχουμε μια θετική προσέγγιση με κάποια σχόλια, σημαντικά θα έλεγα. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην Κομισιόν πως η διαφάνεια των τιμών της πρέπει να βελτιωθεί. Θεωρώ πως ε, το επαρκές ε, σύστημα προστατεύει υπερβολικά τα εμπορικά μυστικά και έτσι οι εταιρείε δεν αποκαλύπτουν ε, δεδομένα στους καταναλωτές και στο κοινό. Γενικά συμφωνώ με αυτά τα οποία προτείνει η εισηγήτρια όσον αφορά τα διάφορα τμήματα του κόστους, αλλά πρέπει να είναι ακόμη πιο διάφορα να περιέχει, π.χ. το κόστος ε, της ε, διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων. Επίσης πρέπει να διαχωριστούν οι πτυχές εκείνες οι οποίες αφορούν την αναδιάρθρωση ε, του άνθρακα. τώρα μπαίνουν όλα μαζί, αλλά θεωρώ πως το πυρηνικό κομμάτι και το κομμάτι των ορεκτών είναι τελείως διαφορετικά και πρέπει να τα αναφέρουμε διαφορετικά. Επίσης, συμφωνώ με την ανάγκη η Κομισιόν να εγκρίνει τη μεθοδολογία ανάλυσης των κρατών μελών, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές, έτσι ώστε να είναι όντως συγκρίσιμα και λεπτομερή τα δεδομένα στα κράτη-μέλη. Επιπλέον, η εισηγήτρια λέει πως για λόγους ποιότητας των δεδομένων μόνο οι καταναλωτές μπορούν να διακριθούν μόνο σε νοικοκυριά και μη νοικοκυριά. Πρέπει να πω πως εδώ πέρα δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πρέπει να υπάρχουν δεδομένα για διάφορους τύπους καταναλωτών. Βιομηχανία έντασης ενέργειας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λοιπούς βιομηχανικούς καταναλωτές για να δούμε πού βρίσκεται το κόστος και πώς επηρεάζονται οι διάφοροι καταναλωτές από τις τιμές. Τέλος, υπάρχουν κάποια κρυμμένα κόστη όπως οι φοροαπαλλαγές, παρεκκλήσεις, λοιπές ενισχύσεις από τα κράτη-μέλη τα οποία δεν τα αναφέρουμε στην πρόταση παρά το ότι θα έχουν μεγάλη σημασία για την διαφάνεια και για να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα για να δούμε το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Συνολικά μπορώ να πω πως α, βεβαίως θα καταθέσω τροπολογίες σύμφωνα με τα όσα ανέφερα περίπου και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους κοιόδης ε, συνεισηγητές όπως ε, μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκιώδη Σιγητά. Από τους φιλελεύθερους, ο κύριος Φιλίπ Ντεμπάκερ. Καταλαβαίνω γιατί δεν με βρίσκεται, γιατί δεν έχω το καρτελάκι μπροστά μου. Τώρα θα εκπροσωπήσω τον κύριο Τερέσκα, δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Θεωρεί ότι δεν είναι επίμαχο το θέμα, δηλαδή ήδη έχει εφαρμοστεί από πολλά κράτη-μέλη. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν σαφείς κατηγορίες για συλλογή δεδομένων εδώ. Τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη, ε, συλλέγουν φόρους, ε, υπάρχει το στοιχείο του κόστους που αφορά τι ανανεώσιμε, αλλά όχι. Βασικά είναι μη συγκρίσιμα τα δεδομένα. Αυτό είναι προβληματικό, γιατί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρειάζονται στατιστικέ για να βασίσουν πάνω σε αυτέ τι πολιτικέ του. Θα πρέπει λοιπόν η ποιότητα των δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη να είναι στο σωστό επίπεδο. Θα πρέπει να κάνουμε επίση ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων, ούτω ώστε ε, να μην συγκρίνουμε δεδομένα ας πούμε, από νοικοκυριά και από βιομηχανικού χρήστε, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση οι συλλογές δεδομένων της Eurostat, ε, η πρόταση της Κομισιόν θέλει απλώς να νομιμοποιήσει αυτή την πρακτική που γινόταν σε θελοντική βάση. Για το σχέδιο γνωμοδότησης, τώρα πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Τρίσκα ε, χαιρετίζει την έφαση ε, στην καλύτερη νομοθεσία, σε επιστημονικά δεδομένα και στην ε, δια, διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία και για να προστατεύσουμε τις, την εμπιστευτικότητα ε, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποια πράγματα ο εισηγητής, ε, πώς θα προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις και πώς θα έχουμε από την άλλη σαφή και ευκρινή δεδομένα. Ευχαριστώ. Από, τους... από την ΚΟΕ, η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση εξ ονόματο του Σκιώδου Συγητή τη ομάδα μου, του κύριου Σιλικιώτη, ο οποίο συμμετέχει αυτή τη στιγμή στην Εξεταστική Επιτροπή για την Εκπομπή Ρήχων στην Αυτοβιομηχανία. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές που χρεώνονται στους οικιακούς καταναλωτές για το φυσικό αέριο αλλά και για την ηλεκτρική ενέργεια. Απότερος μας στόχος είναι να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά από την εσχροκέρδεια, να διασφαλίσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και να επιτύχουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των νοικοκυριών με όσο το δυνατό πιο χαμηλές τιμές. Οι τροπολογίε που θα καταθέσουμε στοχεύουν στο να ενισχυθούν οι συνιστώσει ανάλυση ώστε να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα η οποία να αντανακλά την πραγματικότητα για τι τιμέ που χρεώνται στα, στα κράτη-μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό όμω, θεωρούμε, πω είναι τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν άμεσα στην διόρθωση τη μεθοδολογία αναφορικά με τον έλεγχο των τιμών και οι αρμόδιε υπηρεσίε να εντατικοποιήσουν του ελέγχου που διενεργούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, colleague. Now I would like to ask some comments. Κάποια σχόλια τώρα από τον εκπρόσωπο της Eurostat και από τη Γενική Διεύθυνση Stat. Okay, thank you, Mr. Chairman, dear members of the European... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, η ενέργεια είναι μία από τι δέκα βασικέ προτεραιότητε τη Κομισιόν υπό την Προεδρία του Γιούνκερ. Το πακέτο τη Ενεργειακή Ένωση έχει τρει πρωτοβουλίε Κομισιόν. Η μία είναι ένα πλαίσιο για στρατηγική, ούτω ώστε να έχουμε μία ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση ε, με ουσιαστική συνιστόση για το κλίμα. Ε, ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της διαφάνειας ενεργειακής αγοράς. Λεπτομερή δεδομένα, απαραίτητες πληροφορίες που να βασίζονται σε στοιχεία για να φτιάξουμε σοβαρή πολιτική και να υπάρξει απόλυτη ενσωμάτωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και ανθεκτικότητα της Ενεργειακής Ένωσης. Το Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι η Eurostat, συλλέγει πληροφορίες για τις ε, τιμές ενέργειας εδώ και πέντε δεκαετίες. Το 1990 μια ε, οδηγία του Συμβουλίου τέθηκε σε ισχύ που μιλάει για τη μεθοδολογία για τη συλλογή των τιμών ε, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για τους βιομηχανικούς χρήστες. Για τα νοικοκυριά ε, γίνεται η συλλογή αυτών των δεδομένων σε εθελοντική όμως βάση. Τα τελευταία ένα-δύο χρόνια η Κομισιόν έχει λάβει κάποια ανησυχητικά μηνύματα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συλλογή των δεδομένων των τιμών ενέργειας για τα νοικοκυριά κινδύνευε λόγω της έλλειψης ε, νομοθεσίας. Είναι σαφές ότι η συλλογή των δεδομένων γίνεται σε θελοντική βάση και όταν οι πόροι δεν επαρκούν, θα σταματήσει να γίνεται απλούστατα. Δεν θα εκπλήσει κανένα σας ότι η Κομισιόν αποφάσισε να αντιδράσει για να εγγυηθεί τη συνέχιση της ε, συλλογής δεδομένων για το φυσικό αέριο και το, το ηλεκτρικό ρεύμα. Η πρόταση, ε, το σχέδιο πρότασης συζητήθηκε πάνω από ένα χρόνο με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη για να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των δεδομένων, εξασφαλίζονταν και την τεχνική συγκρισιμότητα και την επαρκή ορατότητα. Θέλουμε μια μεθοδολογία που θα εγγυάται ενιαία, ενιαία και το υπογραμμίζω, ε, αναφορά των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πιο σημαντικό, η πρόταση εφαρμόζεται με όλες τις αρχές και τις νομικές εγγύησεις που προβλέπει το Στατιστικό Γραφείο Πληροφοριών και το, ο 223. Αυτό είναι το πλαίσιο ε, για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι στατιστικές θα πρέπει να γίνονται με βάση την αρχή της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας κόστους κόστους-οφέλους, της μείωσης του άχθους της διοικήσης και στους ε, ιδιώτες, προστατεύοντας όμως ε, τη στατιστική εμπιστευτικότητα. Είναι σαφές ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Μπάρμπαρα κάπου την εισηγήτρια, καθώς και τους κοιόδης εισηγητές για τη δουλειά που κάνουν και τους συμβούλους τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε για την πρόταση αυτή. Uh, και προθεσμία για αποβολή τροπολογιών η 13η Απριλίου έτους 2016, 12 ώρα το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Ήτρε 24 Μαΐου ψηφοφορία στην Ολομέλεια πιθανότατα ένα μήνα μετά. Επόμενο σημείο. Έκθεση πρόοδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείο 14. Η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο είναι η συγγήτρια. Να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση προόδου αυτή είναι πολύ επικαιρή. Αναμένεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το τέλος του έτους. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Ήτρε. Διεξήχθη στις 17 Μαρτίου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η ΕΝΒΗ, σύμφωνα με το άρθρο 54 συμμετέχει και αυτή στις διεργασίες με αποκλειστικέ αρμοδιότητες για τα κριτήρια βιωσιμότητας, για τα βιοκαύσιμα. Άρθρο 54. Αποκλειστική αρμοδιότητα για κριτήρια βιωσιμότητας. Αποκλειστική αρμοδιότητα. Η υπόλοιπη έκθεση συντάσσεται βάσει του άρθρου 53 συν. Η κυρία Λόπεθ Μπερμέρο, αν έχει την καλοσύνη να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις υπενθυμίσεις, σας ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που είστε παρόντες, όσοι είστε δεδομένης της ώρας που είναι, δεδομένων των συνθήκων στι οποίε ε, βρισκόμαστε. Θα ήθελα καταρχά να δώσω έμφαση σε κάποιες πτυχές που θεωρώ σημαντικές και που βρίσκουν σύμφωνα στις περισσότερες ε, πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε κάποια από τα θέματα που θα θέλαμε όμως να πάμε λίγο πιο μακριά στην έκθεση και που θα, ε, τα δουλέψουμε και με τις τροπολογίες. Πρώτον, μια μεγαλ, ένας μεγαλύτερος ορισμός Τη σημασία του τοπικού παράγοντα και το να έχουμε αστικές πολιτικές επάρκειες, παραγωγή και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος σε συλλογικό επίπεδο. Υπάρχει μια τάση ε, νέων φαινομένων, η αυτοκατανάλωση και η αυτοπαραγωγή. Εμείς φυσικά τα υπερασπιζόμαστε αυτά τα φαινόμενα, ε, ειδικά απέναντι σε κάποιες κυβερνήσεις όπως της Ισπανίας. Το δικαίωμα να συμμετέχεις στην παραγωγή και στη διανομή της ε, ηλεκτρικής ενέργειας ως μικρός παραγωγός. Αλλά είναι πιο εύκολο να υπάρξει μια ενσωμάτωση, να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής που θα στοιχηματίζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, δεύτερον, οι στόχοι για το 2020-2030. Στην έκθεση ξεκαθαρίσαμε ότι θέλουμε οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο να διατηρηθούν. Θέλουμε όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι ο ορίζοντας ε, αυτός του 2020 2030, ε, ενώ κρατάει τα, την παραγωγή ενέργειας και από τα ορυκτά καύσιμα σε αυτή τη δεκαετία, θα πρέπει μέχρι το 50 να, τα έχει, να έχει στραφεί αποκλειστικά στις ανανεώσιμες. Το 40% είναι απόλυτα ε, εφικτό στόχο σε εθνικό επίπεδο για αυτό το χρονικό ορίζοντα και θα πρέπει να συνεισφέρει σε ένα υψηλότερο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, για τις χώρες που δεν τα καταφέρνουν. Δεν θέλουμε να τις τηλητεύσουμε. Θέλουμε απλώς να τονίσουμε τις ε, πολιτικές που δεν λειτουργούν. Κάτι σημαίνει να καταγγείλουμε την ε, διάλυση αναδρομικά του συστήματος ε, βοήθειας που υπήρχε. Η πολιτική επίσης ανταγωνισμού θα έπρεπε να είναι πιο ε, για να διορθώσει τα λάθη. Όταν έχουμε από τη μία μεγάλες ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ρυθμιστικές αρχές που υπάρχουν, έχουν μια συμπεγνία μεταξύ τους. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο κυρίαρχο, δημοκρατικό και βιώσιμο. Κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμο. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθορίσουμε με την ε, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τη μετάβαση προς αυτό το νέο μοντέλο που θα είναι κοινωνικά βιώσιμο και παραγωγικά αποτελεσματικό. Θέλω να τονίσω ε, ότι πρέπει να υπάρχουν εθνικά σχέδια και να εκπονηθούν με σοβαρότητα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για τη συνεργασία σα και να σα εκφράσω το ενδιαφέρον μου για να συντάξουμε τροπολογίε μέσα στι προβλεπόμενε προθεσμίες. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Σκιώδη συζητητή για το ΕΛΚ, ο συνάδελφο Μπένσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο εκθέσεώς της. Είναι σαφές από αυτήν ότι συμφωνούμε επί ενός θεμελιώδου στοιχείου. Η Ευρώπη πρέπει να ηγείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό είναι σημαντικό. Να ξεκαθαρίσω ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αποτελεσματικός τρόπος να μειώσουμε την εξάρτηση επί των ορυκτών καυσίμων και θα δημιουργήσουμε έτσι μια οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακο. Οι ανανεώσιμε συμβάλλουν τα μάλα στη βιωσιμότητα. στι εξαγωγέ ανάπτυξη, επασχολημότητα, έρευνα και καινοτομία. Γι' αυτό πάνω σε αυτό η και εγώ θα συμφωνήσουμε. Πέραν αυτού, φοβούμαι ότι η συγγήτρια λησμόνει σε κάποια κρίσιμα σημεία στο σχέδιο εκθέσεως. Η συγγήτρια θα ήθελε να επικρίνει την πρόοδο που έχει γίνει προς τους στόχους του 2020. Εγώ αυτό το επικροτώ. Είμαστε καθοδόν προς την επίτευξη του στόχου του 20%. 25 από τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αναμένεται να πετύχουν τους στόχους του 2020 και 19 από αυτές θα ξεπεράσουν τους στόχους. Η συγγήτρια θα ήθελε να κατονομάσει τις χώρες που πρέπει να κάνουν και άλλες προσπάθειες. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το πώς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φτάσουν εκεί. Μπορούν η συγγήτρια θέλει να χρησιμοποιήσει την έκθεση για να αντιμετωπίσει εθνικά ζητήματα. Για την ώρα, εγώ βλέπω διάφορες παραπομπές σε θέματα που αφορούν ισπανικά συμφέροντα. Και για να συμφωνήσουμε στην έκθεση, θα πρέπει η έκθεση να παραμείνει εντός θέματος. Ήδη επέσα την προσοχή της ηγήτριας σε κάποιες βασικές πτυχές για τους σκοπούς της εκθέσεως. Πιο πρόσφατα, στην τελευταία συνεδρίαση Ήτρε, Αυτές οι βασικές πτυχές φαίνεται ότι δεν συμπεριλήφθησαν στο σχέδιο εκθέσεως τελικά. Γι' αυτό να τονίσω κάποιες βασικές προτεραιότητες του ΕΛΚ εκ νέου. Επίσης θα είναι θέματα τα, για τα οποία θα υποβάλουμε τροπολογίες. Για το ΕΛΚ είναι εξίσου σημαντικό η έκθεση να δηλώνει σαφώς ότι οι εθνικές αρμοδιότητες για το ενεργειακό μείγμα θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Σαφής προτεραιότητα για την ανάπτυξη των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας είναι η σωστή ανάλυση του κόστους και να αναπτυχθεί και η αγορά η σχετική για αυτές τις πηγές ενέργειας. Θα συμφωνήσει η με μένα, διότι είναι κάτι σημαντικό για την τιμολόγηση της ενέργειας στην Ευρώπη, για τους καταναλωτές και στο τέλος, τέλος για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο, στη σχέση κόστους απόδοσης και στην ανταγωνιστικότητα των ανεωσίμων πηγών ενέργειας, στην ενεργειακή στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Και θα πρέπει να υπάρχουν και προοπτικές για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες, τους στόχους που έχουν θέσει για θέρμανση και ψήξη. Δεν αντιμετωπίζονται σωστά τα θέματα στην έκθεση για την ώρα. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο συνεχιζόμενο έργο του Κοινοβουλίου για τη στρατηγική για θέρμανση και ψήξη και ε, το έργο που επικείται για την αφαίρεση του άνθρακος, για τη μείωση της κατανάλωσης άνθρακος εκπομπών άνθρακος. Προσβλέπω λοιπόν στη συνέχιση των συζητήσεων με την εισηγήτρια και με τους σκιώδεις εισηγητές τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφε λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μόλναρ, εισηγητής για το S&D. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε την για την έξοχη δουλειά που έκανε. Είναι πολύ καλή βάση αυτή για περαιτέρω πρόοδο, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα είναι ισορροπημένη. Η μεθοδολογία και η γενική προσέγγιση που ακολούθησε η εισηγήτρια σύμφωνα με την οποία οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας δεν αφορούν μόνο την προστασία του περιβάλλοντος και δεν είναι μόνο θέμα πρασινίσματος, αλλά είναι σημαντικό να δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας ποιότητας και να αναπτυχθεί η τεχνολογία, η υψηλή τεχνολογία, προθυμένη τεχνολογία στην οικονομία και να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης, η ενεργειακή εξάρτησή της. Αυτή είναι στόχη μας και είναι πρόσδεκτη η προσέγγιση της. Συμφωνούμε επίσης με την εισηγήτρια ότι ένα σημαντικό ποσοστό των κρατών μελών θα πετύχει τους στόχους του 2020. Θα πρέπει να ονομάσουμε, να κατονομάσουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι προοδευτικές και εκείνες που υστερούν, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου χώρας, δυστυχώς της Ουγγαρίας, η οποία δεν αποδίδει καλά. Έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες όσον αφορά αυτές, να τονίσω μόνο δύο σημαντικά ζητήματα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά αποκλίνους, απόκληση απόψεων μεταξύ ημών και του ΕΛΚ που πιστεύουν ότι κατά την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να διατηρήσουμε τα στοιχεία του στόχου, τους δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο λόγος για την καλή πρόοδο κατά το παρελθόν ήταν οι στόχοι που είχαν τεθεί, που ήταν δεσμευτικοί στόχοι και συγκεκριμένοι στόχοι για τα 28 κράτη-μέλη. Ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό και μετά το 2020, αφού πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε, δηλαδή ε, τον... και θεωρούμε ότι ο στόχος που έχει τεθεί το 27% δεν είναι αρκετά φιλόδοξος. Εν πάση περιπτώσει χρειάζονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι και έχουμε υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Εν γέννη πρέπει να είναι ξεκάθαρο στην έκθεση ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το διοικητικό άχθος και την γραφειοκρατία και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, διότι αυτά αποτελούν εμπόδια για την διάδοση της χρήσεως των ανεωσίμων πηγών ε, ενέργειας. Υπάρχουν διάφοροι δασμοί στα κρατη και φόροι για προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι πολύ παράδοξη κατάσταση και εκείνοι που παράγουν τα προϊόντα και οι πελάτες θα πρέπει να υπερκεράσουν τις επαχθείς αυτές διαδικασίες που αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη των στόχων στο μέλλον. Στο τέλος να σας πω κάτι, μια πρόταση έχω, συμβολικής αξίας ενδεχομένω. Λοιπόν, οι πολιτικοί προσπαθούν να δώσουν παραδείγματα, να, να γίνουν παραδείγματα με τον τρόπο ζωής τους. Στο Λευκό Οίκο, στη Ουάσιγκτον Φερρυπίν, υπάρχουν ηλιοθερμοσυσσωρευτές στη στέγη. Ε, και στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ανεμογεννήτριες. Θα πρέπει να δώσουμε και εδώ στις Βρυξέλλες το παράδειγμα, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να δώσουμε το παράδειγμα ότι θερμαίνονται ή ψύχονται οι καταστάσεις του Κοινοβουλίου ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι κάτι συμβολικό, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται τέτοια απτά σύμβολα για να τα απευθύνουμε στους πολίτες μας. Και νομίζω ότι στο τέλος, όσον αφορά την έκθεση, θα πετύχουμε έναν καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε, για τα σχόλιά σας. Η κυρία Βανμποσιούτ έχει το λόγο. συγκήτρια του ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχεδόν το πετύχατε. Μπράβο. Ναι, ναι, είναι η δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά, αν περιμένετε λίγο, θα το πετύχω. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντίδρασή μας για την έκθεση πρόοδου νομίζω πως ε, είναι αναμενόμενη καθώς περιμέναμε αυτή την έκθεση. Είναι θετικό το ότι όλα τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο για να πετύχουν τους στόχους του 2020 και βλέπουμε εδώ πέρα πως ε, πρέπει να δούμε τις ανανεώσιμες πηγές ως ένα οικοσύστημα από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή πρέπει να έχουμε μια αγορά ενέργειας η οποία θα λειτουργεί σωστά. και βλέπουμε πως ε, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να φέρουμε. Πρώτα απ' όλα η εισηγήτρια μας λέει πως ε, Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία πλέον δεν βασίζονται στην ε, τρέχουσα κατάσταση στα κράτη-μέλη και εδώ πέρα θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Ένα άλλο θέμα είναι πως ε, θέλει σε όλες τις συμφωνίες εδώ πέρα η συγγήτρια να εμπλέξει τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Εντάξει, μπορεί να είναι σημαντικό αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες. Γιατί να περιληφθεί μόνο αυτή η ομάδα και όχι κάποιοι άλλοι. Τρίτο και τελευταίο, πρέπει να γνωρίζουμε πως έχουμε, εργαζόμαστε προς μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και θα πρέπει άρα οι βλαπτικές επιδοτήσεις να καταργηθούν. Και συχνά στην έκθεση μιλάτε για αυστηρούς ελέγχους των τιμών ή για επιδοτήσεις. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πρέπει να αφήσετε την αγορά να λειτουργήσει. Αυτό πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο αυτά και σας ευχαριστώ και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ο Φιλίπ Ντεμπάκερ. πρέπει να πέτυχα και το δικό σας το όνομα. Ε, ναι, ναι, μετά από πέντε φορές. Τελευταία φορά που μιλάω σήμερα. Τώρα αυτή τη φορά είμαι παριστάνω τον κύριο Χερμπράντι. Ξέρουμε πως η κλιματική αλλαγή και οι ανταγωνιστικές ε, τιμές ενέργειας ε, και οι διάφοροι υπάροχοι αποτελούν απειλή για το σύστημα ενέργειας ε, της Ευρώπης και οι ανανεώσιμες πηγές αντιμετωπίζουν κάποια από τα ζητήματα. Ο κύριος Χερμπράντι λοιπόν θεωρεί πως είναι θετικό το ότι η έκθεση τονίζει ότι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν επιτυχάνουν αρκετή πρόοδο για τις ανανεώσιμες φυγές μας ανησυχούν μεταξύ των οποίων το Πενελούξ, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και θεωρούμε πως απαιτείται περισσότερη δράση σε αυτές τις χώρες. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να παραμείνει ηγετική δύναμη στις τεχνολογίες αυτές. Ξέρουμε πως από πέρσι η Ευρώπη πλέον είναι η μεγαλύτερη αγορά ανανεώσιμων και η τελευταία έκθεση του Bloomberg δείχνει πως η Ευρώπη μένει πίσω και στις επενδύσεις οι οποίες έπεσαν κατά 18% κοντά στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, το χαμηλότερο νούμερο από το 2006. Οπότε, για να παραμείνουμε στο προσκήνιο αυτού του αγώνα, ήδη νομίζω πως η Κομισιόν έχει δεσμευτεί ξεκάθαρα και θεωρώ πως τα κράτη-μέλη πρέπει να παραμείνουν προσιλωμένα στο στόχο. Σύμφωνα με τον κύριο Χερμπράντι, η έκθεση προόδου σημαίνει πως ε, αν δεν επιτύχουμε τους στόχους ίσως καταλήξουμε σε εθελοντικούς εθνικούς στόχους οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους επενδυτές να υπάρχει προβλεψιμότητα και ίση όρια ανταγωνισμού. Επίσης πρέπει να τονιστεί η μείωση του κόστους για κάποιες, ε, ενέργειες, για κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια ότι μέτρα μπορούν να ληφθούν περαιτέρω για να μειωθεί το κόστος. Οπότε εδώ πέρα επίσης ε, ξεκαθαρίζουμε ότι σε βάθος χρόνου πρέπει να μπορούν να ανταγωνιστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις ε, παραδοσιακές ε, χωρίς επιδότηση. Επιπλέον τονίζουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας για τη σχετική οδηγία μεταξύ κρατών μελών καθώς έτσι θα αυξηθούν οι επιλογές για συμμόρφωση και το κόστος συμμόρφωσης. Οπότε παρά το ότι η Άλντε υποστηρίζει τα κριτήρια τα αυστηρά για τα βιώσιμα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να θεωρούμε την βιοενέργεια ως ε, επιλογή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Συμπερασματικά λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτές τις ε, νέες τεχνολογίες, αλλά και μια προσέγγιση με βάση την αγορά. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους τώρα, ο σκιώδης ο κύριος Γιάμπορ. Um, ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση, νομίζω όπως είπε και ο Πίκερ η έκθεση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο μια έκθεση πρόοδου ή έκθεση εφαρμογή, θα είναι και η βάση για την αναθεώρηση τη οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και θα πρέπει να θεωρήσουμε την ευκαιρία αυτή για να υποδείξουμε την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε στην αναθεώρηση τη οδηγία αυτή. Με αυτό στο μυαλό, πρέπει να ξεκινήσω με τη δήλωση του Ιούνκερ, που είπε ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο πρώτος παγκόσμιος στις ανανεώσιμες. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος από τους δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Χάνουμε έδαφος στις ανανεώσιμες. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειες μας για να παραμείνουμε ή να ξαναγίνουμε το νούμερο ένα σαν ανανεώσιμες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Να ενσωματώσουμε τους διάφορους κανονισμούς σε ένα πλαίσιο, το, να βάλουμε σε ένα πλαίσιο τα μέτρα των κρατών μελών ε, για την αποθήκευση, για το, τις ρυθμίσεις, για τα δίκτυα κτλ. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα πλαίσιο. Χρειαζόμαστε επίσης μια προσέγγιση με κέρδους καταναλωτές, να ενισχύσουμε τους καταναλωτές ούτως ώστε να γίνουν παραγωγή και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για τις ανανεώσιμες ε, έρευνα, παραγωγή, κατανάλωση και στην ηλεκτρική ενέργεια και στη θέρμανση. Συμφωνώ με το σκιώδη των σοσιαλιστών ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι δεσμευτική εθνική στόχη. Όλα όσα έχουμε τύχει μέχρι στιγμής στην ε, ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες στην Ευρώπη είναι συνέπεια των ε, δεσμευτικών εθνικών στόχων. Μετά το 2020 μας θα τους χάσουμε. Και με ανησυχεί τα μάρλα αυτό, με ανησυχεί η επίπτωση αυτής της εξέλιξης. Επίσης, χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε χρηματοδοτικά συστήματα, τον ορίζοντα 2020, τα διαφορετικά ταμείο συνοχή, το ΕΦΣΙ κτλ θα πρέπει να δώσουν κίνητρα για, τις, ε, για τη χρήση της των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα κράτη-μέλη χρειαζόμαστε εξατομικευμένα μέτρα και μηχανισμούς χρηματοδότησης ανάλογα με το μέγεθος αγοράς, την, ε, τον κίνδυνο των ε, τεχνολογιών, τα διάφορα προφίλ. Επίσης, εξειδικευμένα μέτρα για τους χαμηλόμισθους καταναλωτές για να παρεμποδίσουμε την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη. Και μπορούμε να το πετύχουμε χάρη στις ανανεώσιμες. Επίσης, το καθεστώς πιστοποίησης για τις ανανεώσιμες σε κάθε κράτος μέλος, αυτό το, αναφέρει τον έφερε ο σοσιαλιστής Σκιώδης, αυτός θα πρέπει, αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να παγώσουμε όλους τους φόρους ε, που είναι τεχνική, τεχνική φραγμή για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρειαζόμαστε ε, δεσμευτικά εθνικά ε, σχέδια, ούτως ώστε να έχουμε διαφάνεια, συγκρισιμότητα των σχεδίων για την ενέργεια και για το κλίμα σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, να υπάρχει η προβλεψιμότητα για τους επενδυτές ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξουμε τις υποδομές και τα έργα υποδομών σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουμε να κλειδώσουμε σε τεχνολογίες που δεν είναι κατάλληλες για την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ενεργειακές πολιτικές των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πρέπει να δούμε τις διατομιακές πτυχές. Θα πρέπει να τις ε, ενισχύσουμε. Αναφέρθηκε ότι ο τομέας ψήξη και θέρμανσης είναι βασικό στοιχείο. Εκεί μπορούν να παίξουν πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειαζόμαστε νέα, τα νέα και τα παλιά κτίρια να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες με ανανεώσιμες για ψήξη και θέρμανση. Αλλά πολύ σημαντικό και ο τομέας των μεταφορών. Όχι μόνο να περάσουμε στι ανανεώσιμε ανανεώσιμα καύσιμα στις μεταφορές, αλλά να περάσουμε σε άλλο μοντέλο στο, στις δημόσιες μεταφορές, αλλά και στις ιδιωτικές μεταφορές. Θα υποβάλω και τροπολογία με βάση τα όσα σας είπα και ελπίζω να συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν περιορίζω τις παρεμβάσεις όπως βλέπετε. Ορίστε κυρία μου, έχετε το λόγο. Η κυρία Σπυράκη. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να πω ότι διαπιστώνω ότι η πρότασή της ως βάση για τη συζήτηση έχει πάρα πολλά κενά. Και θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα τη συμφωνία μου με τον ραπορτέρ από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος ε, έδωσε την κατεύθυνση με την οποία συμφωνώ απολύτως. Καταρχήν δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε blame and shame στα κράτη-μέλη. Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι οι εθνικές αρμοδιότητες στο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος θα πρέπει να διαφυλαχθούν και ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν το καλύτερο δυνατό ενεργειακό μείγμα με την καλύτερη δυνατή τιμή. Ως εκ τούτου, οποιασδήποτε αναφορές σε αυστηρούς ελέγχους των τιμών και επιδοτήσεις είναι έξω από το πνεύμα αυτής της κατεύθυνσης. Αντιθέτως, άκουσα και άλλους συναδέλφου να το λένε, θα πρέπει να επιταχύνουμε. Πώς να επιταχύνουμε. Λείπουν από αυτή τη συζήτηση προτάσεις για ενθάρρυνση των δεπενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά στις δημόσιες μεταφορές με βιοκαύσιμα, ως ένας γρήγορος τρόπος για να επιτευχθεί ο αντίστοιχο στόχο, ο οποίο αυτή την ώρα είναι πολύ χαμηλά. Λείπει από την ε, συζήτηση αυτή η παρουσία του EFSI ως εργαλείο χρηματοδότησης ειδικά μετά την δυνατότητα να έχουμε συμπληρωματική χρηματοδότηση στα διαφορετικά ταμεία. Αυτές είναι καταρχήν κάποιες σκέψεις και όσο έχουσα και άλλη ιδιότητα, την ιδιότητα της σκιώδους εισηγητρίας για, την, για το opinion στη Ρέτζη, θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μάριον Ντόναλη, της Γενικής Διευθύνσεως Ενέργειας, η Γενική Διευθύντρια της DG Energy. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις που έκαναν σχόλια. Είναι μια έκθεση που πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Όλες είναι ενδιαφέρουσα, αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μας, διότι ετοιμάζουμε αναθεώρηση της οδηγίας για ανανεώσιμες που πρόκειται να υιοθετηθεί στο τέλος του έτους. Και πρέπει να πούμε ότι θα εμπνευστούμε από το περιεχόμενο αυτής εκθέσεως όταν θα ολοκληρωθεί αυτό. Είναι σημαντικότατο και επικοδομητικό αυτό για μας να έχουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου η ψηφοφορία σας για το 2030 ήταν σημαντικό βήμα και βοηθά το ότι να γνωρίσετε τη σημασία που έχει το σταθερό ρυθμιστικό καθεστώς και ο διάδρομος της ζήτησης που οδηγεί σε μείωση του κόστους τεχνολογίας και μέσω αυτών θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στους Ευρωπαίους καταναλωτές μέσω μειώσεως του κόστους. Κάτι μπορούμε να πετύχουμε να αναθεωρήσω των κειμένων. Είναι πρόσδεκτο επίση ότι το Κοινοβούλιο διευρύνει τι συζητήσει εξετάζει το θέμα ψήξεω και θερμάνσεω που είναι 50% της ενεργειακής κατανάλωσης. Σημαντικότατο οι ανανεώσιμε να παίξουν το ρόλο του εκεί. Παρομοίω τι μεταφορές που ήταν ένας δύσκολο τομέα μέχρι τώρα αλλά εκεί θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο για να κινηθούν προς τα εκεί στο μέλλον. Όσον αφορά κάποιες από τις προτάσεις που ακούστηκαν, καλωσορίζω τα σχόλια που έγιναν όσον αφορά τους καταναλωτές. Οι ανανεώσιμε λόγω της μικρής κλίμακας της τεχνολογίας ανοίγουν την πόρτα προς τη συμμετοχή των καταναλωτών στην ενεργειακή αγορά και αυτό είναι μια τάση ευπρόσδεκτη προς υποστήριξη. Επίσης, καλωσορίζουμε τα σχόλια που κάνατε σχετικά με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι ένας τομέας που θεωρούμε ότι εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε, να επιφέρουμε βελτιώσεις. Με τα χαρά συνεργαστήκαμε γιατί στο κείμενο, αν τα στοιχεία μας είναι κάπως απειρχιωμένα, διότι συνήθως χρησιμοποιούμε στοιχεία Ευρωστάτ που μένουν πίσω δύο χρόνια, αλλά έχουμε και πιο σύγχρονα στοιχεία για το 2015 παραδείγματος χάρη που μπορούμε να τα διαθέσουμε. Βέβαια Εννοώντα ότι δεν είναι μπροστά, αλλά πιο πρόσφατες πληροφορίε. Εν γέννη, Πρόεδρε, δεν θέλω να ακρηγορήσω. ευπρόσδεκτα τα σχόλια που ακούστηκαν, ευπρόσδεκτη η κατεύθυνση τη εκθέσεω. προσβλέπω στο να μα εμπνεύσει αυτή προς το κείμενο που ετοιμάζουμε και αν υπάρχει κάτι με το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε όσον αφορά αριθμού, πληροφορίε κλπ, μην διστάσετε γνωστοποιήστε το μα. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Προθεσμία για αποβολή τροπολογιών 13 Απριλίου 2016 το μεσημέρι. Συζήτηση των τροπολογιών 20 Απριλίου. Ψηφοφορία στην Ήτρε 24 Μαΐου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεύτερη σύνοδος του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ παρόντες είσαστε άκρος υπομονετικοί, σχεδόν εξίσου υπομονετικοί με μένα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τελειώσαμε όλα τα σημεία της συνεδριάσεως στις 20 Απριλίου και 21 Απριλίου θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπής μας το πρωί. Α, Συγγνώμη, η κυρία Συγήτρια, θέλετε να πείτε κάτι. Συγγνώμη, οι προηγούμενοι εισηγητές δεν ήταν καν παρόντες. Ασυνήθιστος εισηγητής είστε για σήμερα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Συγχωρεμένος, Πρόεδρε. Θα κλείσω με εσάς το... τη συνεδρίαση αυτή. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Σας καταλαβαίνω, Πρόεδρε. No, solamente muy brevemente. Πολύ σύντομα. Ναι, εξάλλου. Ξανά ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Άκουσα με προσοχή τις προτάσεις. Όλα όσα είπατε. Άκουσα αυτά που είπε η Κομισιόν. Θα ξαναδούμε τα στοιχεία. Αλλά νομίζουμε ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να αναφερθεί μαζί με τις χώρες ούτω ώστε να δοθούν περισσότερα κίνητρα για να βελτιώσουν οι χώρε τι επιδόσει του στον τομέα των ανανεώσιμων. Ο ρόλο των καταναλωτών είναι πολύ σημαντικό, οι δεσμευτικοί στόχοι. Υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία στι ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια και χάρη σε αυτέ μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Θα πρέπει να υπάρχει επίση ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο χωρί αβεβαιότητε και να υπενθυμίσουμε ότι οι ανανεώσιμες και η δουλειά που κάνουμε εξασφαλίζει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της πράσινης βιομηχανίας, που είναι πρωτοπόρος και που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, όπως είπαν και κάποιοι ισχυώδεις εισηγητές. Τελειώνω. Ξέρω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα φτάσουμε σε συμβιβασμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κλίμα συνεργασίας και Συμφωνώ με τη συμβολική αυτή χειρονομία που πρότεινε ο συνάδελφος. Τη συμμερίζομαι κι εγώ. Και εγώ σα ευχαριστώ κυρία μου. Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά σα. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Και για την Επιτροπή μα και για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συναντηθούμε 20 και 21 Απριλίου. Πρωί-απόγευμα και τις δύο μέρες. Ευχαριστώ.